Mrs. Renate Weber and Mr. De Grandes, and I'll ask them in this order to take the floor. Thank you very Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, μπορώ. Σας ευχαριστώ σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω εδώ για να σας μιλήσω για την αποστολή μας στις προεδρικές εκλογές στο Περού 3 με 7 Ιουνίου, πώς έλαβαν ακριβώς ο χώρο, όχι μόνο ο δεύτερος γύρος των προεδρικών, αλλά και ο πρώτος γύρος και οι κοινοβουλευτικές εκλογές για το Περουβιανό Κογκρέσο. Τολμώ να πω πως ήταν μια επιτυχής αποστολή αυτή των Ευρωπαίων Παρατηρητών. Πρώτον, γιατί η δουλειά που κάναμε εκεί ήταν πολύ σοβαρή. Δεύτερον, επειδή η παρουσία μας εκεί ήταν σημαντική για αυτές τις εκλογές. Και τρίτον, επειδή ακολούθησαν και δραστηριότητες πάνω στις οποίες συνεργαζόμαστε με τους περουβιανούς εταίρους. Η αποστολή αυτή ήταν μια μεγάλη. Φτάσαμε στις 5 Μαρτίου στη χώρα, 10 εμπειρογνώμονες και μερικά από μετά από μερικές εβδομάδες και άλλοι 16 παρατηρητές που αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και θα έμεναν εκεί για πολύ. Επιπλέον, η πλήρης αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έφτασε για τον πρώτο γύρο των εκλογών και βέβαια και για τον δεύτερο. Για τον πρώτο προείδρευε ο συναδέλφος μας Λουίς Τεγκράντε και για το δεύτερο γύρο ο Αγουστίν Τεμέρα. Για πρώτη φορά είχαμε μαζί μας μεταξύ των εμπειρογνωμόνων έναν εμπειρογνώμονα για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας που στην περίπτωση του Περού αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα σας εξηγήσω γιατί σε λίγο. Η δεύτερη σημαντική πτυχή είναι το πόσο μεγάλη σημασία έχει η παρουσία μας εκεί εν ώψη των εκλογών. Και επιμένω πάνω σε αυτό και τολμώ να πω ότι κάναμε τη διαφορά. Η παρουσία μας δηλαδή εκεί έκανε τη διαφορά και θα σας εξηγήσω σύντομα γιατί. Δυστυχώς το Κογκρέσο του Περού δεν προχώρησε σε βαθιά μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος. Ανταυτού αυτό που έκαναν είναι ότι πέρασαν κάποιες τροπολογίες, κάποιες, αφού είχαν ανακοινωθεί εκλογές και αφού ξεκίνησε η προεκλογική διαδικασία. Κάποιες από αυτές που ήταν εννοείται δεσμευτικές, υποχρεωτικές, πρόκειτο για την αρχή που είναι υπεύθυνη για τις εκλογές, που αποφάσισε τις εβδομάδες που ακολούθησαν να αποκλείσει από τις εκλογές κάποιους υποψηφίους, ενώ άλλοι αποσύρθηκαν από τις εκλογές επειδή θέλησαν να προστατεύσουν την νομική οντότητα του κόμματός τους. Οπότε στο τέλος από τους 19 υποψήφιους στην Προεδρία μόνο 10 παρέμειναν ε, στην εκστρατεία αυτή και βέβαια με πολλή αβεβαιότητα μέχρι μάλιστα την τελευταία μέρα πριν τις εκλογές, όπου δεν γνωρίζαμε στα σίγουρα ποιος άλλος τελικά θα αποσυρθεί. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Συγχρόνως, στα μέσα ενημέρωσης, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξαν διάφορα άρθρα, τα οποία αμφισβητούσαν ε, την δυνατότητα της χώρας να οργανώσουν δημοκρατικά τις εκλογές αυτές. Και σχολίαζαν τη δυνατότητα υποψηφίων να είναι υποψήφοι και κατά πόσο το γεγονός αυτό, η συμμετοχή τους δηλαδή στην εκστρατεία, πώς θα επηρέαζε την εκλογική διαδικασία. Πάντως, όντας εκεί και συζητώντας με όλες τις αρχές, εποφελούμενη 100% διαφάνεια από πλευρά των Περουβιανών, γιατί είναι αλήθεια ότι είχαμε πρόσβαση στα πάντα, σε ό,τι θέλαμε, χωρίς κανένα εμπόδιο. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα, μετά από σοβαρή νομική ανάλυση του εκλογικού περιβάλλοντος, ότι όλα όσα έγιναν, όσο και αν αμφισβητούνται από πλευράς του δικαιώματο κάποιου να είναι υποψήφιος ή όχι, ε, παρόλα αυτά όλα βασίζονταν στην νομοθεσία, που μπορεί να μην ήταν πάντα καλή, αλλά βασίζονταν στην νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του συντάγματος. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για πάτη, για παραπλάνηση. Δεν υπήρξαν πολιτικές πιέσεις από τους οργανωτές των εκλογών. Και από τη στιγμή λοιπόν που αντιληφθήκαμε ότι αυτή ήταν η πραγματικότητα, το είπαμε και το επαναλάβαμε αυτό ξανά και ξανά. Όσον αφορά λοιπόν, αυτά ήταν τον πρώτο γύρο για τις προεδρικές εκλογές και για το Κογκρέσο. Οι συζητήσεις έγιναν για αυτά τα διαδικαστικά ζητήματα και όχι τόσο για το μέλλον της χώρας. Παρόλα αυτά, οι εκλογές έγιναν. Οργανώθηκαν καλά. Όλα όσα έγιναν την ημέρα των εκλογών έγιναν καλά και όλοι δέχτηκαν και τα αποτελέσματα. Ο δεύτερος γύρος ήταν πιο εύκολος. Πάλι ήταν μια έντονη συζήτηση αυτή που έγινε μεταξύ των υποψηφίων και είναι ενδιαφέρον εδώ να αναφέρουμε ότι η κυρία Κέκο Φουτσιμόρη ήταν η επικρατέστερη με 42.000 διαφορά ψήφων. Δέχτηκε όμω τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι τα καταφέρνει κάπω καλύτερα το Περού από η Αυστρία, γιατί το Περού δεν ζήτησε να ξαναγίνουν οι εκλογέ επειδή η διαφορά είναι τόσο μικρή. Ο κύριος Πέντρο Κουτσίνσκι τελικά κέρδισε τις εκλογές με αυτή τη διαφορά 42.000 ψήφων από την Βουτσιμόρη. Πολύ δημοκρατικά έγιναν ε, οι εκλογές και όταν ο κόσμος περίμενε τα επίσημα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακό να δούμε πόσο καλά έγιναν όλα και πώς τα μέλη των διαφέρων κομμάτων και ψηφοφόροι συμπεριφέρθηκαν. Οπότε ο κύριος Κουτσίνσκι τέλη Ιουλίου θα αναλάβει ως νέος πρόεδρος του Περού. Θέλω επίσης να αναφέρω και τι έγινε στη συνέχεια και με αυτό θα σταματήσω. Οι δραστηριότητες που ακολούθησαν θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικές στην περίπτωση του Περού. Διότι αποτελούν μια μεγάλη επιτυχία του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάσει τις δημοκρατικές εξελίξεις σε μια χώρα. Την επόμενη εβδομάδα έτσι κι θα επιστρέψω και πάλι στο Περού για να παρουσιάσω την τελική μας έκθεση και τις συστάσεις μας, αλλά επιπλέον έχουν αρχίσει κάποιες δραστηριότητες που έχουμε σκεφτεί και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέρφους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί και πρόθυμοι να συνεργαστούν με τα μέλη του Κογκρέσου. Αλλά αυτό που επίσης μπορώ να σας πω ότι εγκρίθηκε η συνεργασία με το Κογκρέσο του Περού, οπότε ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και τα επόμενα χρόνια. Σταματάω εδώ και αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρος. Ο ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Και εγώ να επαναλάβω τα συγχαρητήρια για την νίκη του Ιουνίου στις, στις 5 Ιουνίου που νίκησε ο κύριος Κοτσίνσκι και επίσης πιστεύω ότι άξιζε ε, να κερδίσει η εργασία όσον αφορά τις εκλογές ήταν πάρα πολύ αξιόλογη. Πρώτος και δεύτερος γύρος για τις προεδρικές και τις κοινωνικές εκλογές. Συμφωνώ με όλα όσα ακούσαμε σήμερα. Με όλα σας τα συμπεράσματα και παρατηρήσεις. γιατί πρόκειται για κάποια κατάσταση την οποία παρακολουθήσαμε από κοντά που είχε μεγάλη ε, σημασία, ήταν πολύ σημαντικέ αυτές οι εκλογές. Έχουμε εδώ ως πρόεδρος των σχέσεων με τις ε, χώρες των Άνδιων και του Συμφώνου των Άνδιων αλλά θα πρέπει να συγχαρούμε και τον πρόεδρο της, ε, των παρατηρητών της, των εκλογών της 10ης Απριλίου. Νομίζω ότι επέδειξε ο λαός του Περού δημοκρατική, υποδειγματική συμπεριφορά και οριμότητα δημοκρατική. Οπότε και ο ΟΜΠΕ, ο Οργανισμός για τις Εκλογές, ε, επίσης και οι επιμέρους εκλογικές επιτροπές επέδειξαν επίσης το σωστό επαγγελματικό πνεύμα. Βλέπουμε τώρα τι σχέσεις υπάρχουν μεταξύ Ευρωπαϊκής και Περού και γι' αυτό και έχουμε πολύ καλή λειτουργία της εμπορικής συμφωνίας που ισχύει εδώ και δύο χρόνια και προσφέρει πολλές δυνατότητες τόσο ώστε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο και οι δύο πλευρές τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από αυτή την εμπορική σχέση. Επίσης είπαμε ότι προσωρινά ισχύει η συμφωνία για τη βίζα του διαβατηρίου για την σύντομη διαμονή των ε, Περουβιανών στον χώρο του Σέγγεν. Για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία ήταν σημαντικό ρόλο του Κοινοβουλίου. Και τώρα και κάτι άλλο το οποίο αφορά το παρελθόν. Αλλά είναι κάτι το οποίο η κυρία Βέμπερ το ετώνησε και αυτή, ότι πρόκειται για μια εξαίσια ευκαιρία, ούτως ώστε ε, ε να μπορέσουμε μέσω του κύρους των ε, ε, αυτών που έχουν λάβει τις επαφές να συσφίξουν τις σχέσεις μας με το Πέρο γιατί έχουμε τον καινούριο πρόεδρο και έχουμε και ένα καινούριο κογκρέσο. Αλλά βέβαια ο Φουχιμόρη εκεί έχει την ε, πλειοψηφία. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται και κατανόηση. Το δέχονται αυτό οι συνομιλητές μας και δέχονται την διαμεσολάβησή μας. Οπότε έχουν ξεκινήσει σχέσεις τέτοιου είδους που έρχονται εδώ αυτοί οι, ε, οι εκπρόσωποι αυτού του προεθνικού κινήματος και έρχονται και λένε ότι και από τις επαφές μαζί μας κάπως μαθαίνουν και επίση αναζητούνται διέξοδοι και λύσεις σε κοινά προβλήματα. Πρόκειται για κάτι που προσφέρεται να εκμεταλλευτούμε και δεν είναι θεωρητικό το θέμα, είναι πρακτικό και αφορά αυτή την σπουδαία χώρα που προοδεύει και εξυγχρονίζεται και που έχει πάρα πολύ σημαντική γεωστατική θέση στην Νότια Αμερική. Πά, πρόεδρε, πρόεδρε, κάτι άλλο που θα ήθελα να σα πω. Γιατί εδώ έχουμε τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βαλκάρθα, τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου. Θα λάβει και αυτό βέβαια το λόγο. Θέλω να πω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ω χειρονομία η πρόκληση τη 28η ε, Ιουλίου. Ε, και εκεί θα μα εκπροσωπήσει στην πρόσκληση που έχουμε κάνει προ την άλλη πλευρά. Εκεί θα μα εκπροσωπήσει και τον ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα πρώτου δώσω το λόγο στους δύο συναδέλφου, οι οποίοι ζήτησαν το λόγο θέλω να χαιρετήσω την παρουσία εδώ μιας ε, αντιπροσωπείας από βουλευτές του Πακιστάν που είναι παρόντες εδώ μαζί μας. Θα τους ε, παρακαλούσα, προσκαλούσα να ακούσουν τη συνεργασία συνεδρίασή μας στο κανάλι 2 τα αγγλικά. Ο κύριος Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους παρατηρητές, αυτούς οι οποίοι ήταν παρόντες και τους... Ε, εμείς έχουμε παρακολουθήσει από πολύ κοντά τις ε, εκλογές γιατί είχαν πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο για το Περού αλλά για όλη την Αμερικανική Ήπειρο. Θέλω να προσθέσω και ορισμένες σκέψεις εδώ έχοντας ακούσει αυτά είπε ο κύριος, η κυρία Βέμπερ και ο κύριος Δεγράντες, ε, Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Κουτσίνσκι θα έχει δυσκολίες για να μπορέσει να διαχειριστεί τη χώρα αυτή όταν έχει μια πλειοψηφία εναντίον του στο Κογκρέσο του Περού και γνωρίζοντας ότι δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει όλες τις ψήφους εναντίον της ε, Φουχιμόρη και κάποιες από τις ψήφους που πήρε μπορεί να τις θεωρήσουμε δανεικές ουσιαστικά. Ε, υπήρξε αυτό το, το μέτωπο το οποίο τον υποστήριξε, το ευρύ μέτωπο, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσει να τον υποστηρίζει και στο μέλλον. Αυτό είναι μια από τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει στη χώρα αυτή και έχει δύο σημαντικές ε, προκλήσεις. Το ένα είναι το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης, όπως ανέφερε ο Ντεγκράντε και εκεί η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά για να βοηθήσει αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπίσει την εξορρυκτική βιομηχανία και φυσικά όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά, το λαθεμπόριο ναρκωτικών κτλ. Και ένα δεύτερο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό είναι γιατί έχει τόσο μεγάλη δύναμη ο φουχημορισμό, όπω θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε. Και για μένα το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αρκετά εδρεωμένο το, το σύστημα των κομμάτων δεν είναι αρκετά δομημένο ώστε να επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν, ε, να υπάρξουν κατευθύνσεις που να ανταποκρίνονται στις αιτήσει των εκλογέων. Το γεγονός ότι αναδύονται και εξαφανίζονται πολλά κόμματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η περίπτωση του Φουχημόρη και της κόρης του είναι χαρακτηριστική. Αυτό το λέω γιατί μπορεί να είναι κάπως ντεμοντέ αυτό ότι να το λέει κανείς ότι τον έχουμε ένα ισχυρό κομματικό σύστημα αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και στην περίπτωση του Περού έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ακριβώς έτσι αλλά το να υπάρξει ένα σταθερό κομματικό σύστημα σε μακροχρόνιο επίπεδο θα ανταποκριθεί και στις αιτήσεις των εκλογέων αλλά και θα εξασφαλίσει και τη σταθερότητα. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Η κυρία Βιλβάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, πρέπει προφανώς να ευχαριστήσω τη Ρενάτε για το εξαιρετικό της έργο και τον Λουίς Τεγκράντες από την πλευρά της αντιπροσωπείας λοιπόν του Κοινοβουλίου, αυτά τα δύο άτομα. Εγώ θα ήθελα να διατυπώσω το εξής ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τις εκλογικές μετατοπίσεις οι οποίες εμπόδισαν να, μάλλον επέτρεψαν την εκλογή κάποιων υποψηφίων έχουν κατανοήσει τα πολιτικά κόμματα ότι χρειάζεται να υπάρξει μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου εν ώψη των ε, ε, επομένων εκλογών. Υπήρξαν κάποιες ε, αντιπαραθέσεις, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι κάποιοι υποψήφοι αποκλείστηκαν, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το, είχαμε, το είχαν υπολογίσει πολύ, αλλά είναι και απόρρια αυτή τη νομοθεσία. Μήπω λοιπόν θα είναι απαραίτητε κάποιε μεταρρυθμίσει στο εκλογικό δίκαιο για να, για να αποτραπούν τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Και δεύτερον, θα ήθελα να ξέρω αν κατά την άποψή σα κάποιοι από του υποψήφιου που δεν είχαν τη δυνατότητα να ε, διαγωνιστούν για την Προεδρία, αν θα μπορούσαν να έχουν μια δυνατότητα να ανταγωνιστούν την Φοχημόρη. Αν θα μπορούσαν λοιπόν, από ό,τι είδαμε, ε, θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο θα υπήρχαν και δυνατότητες να υπάρχει μια ευρύτερη παρουσία υποψηφίων. Ο κύριος Σεμπαστιά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή που μας επέτρεψε να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτήν την αντιπροσωπεία και μας προσκάλεσε να έρθουμε και εδώ. Ευχαριστώ και την πρόεδρο της αντιπροσωπείας για τα λόγια της και τον Λουίς Δεγκράντες. Η αντιπροσωπεία πολύ συγκεκριμένα έφερε σε πέρα στην αποστολή της. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι δηλώσεις που έγιναν εκεί οι επίσημες τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Υποπιτροπής ας πούμε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ε, σαφείς και είχαν ιδιαίτερη αξία. Αναγνωρίσαμε ότι εργαστήκαμε με κάθε διαφάνεια και με την κάθε καλή βούληση από κάθε πλευρά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, υπήρχε πλήρης διαφάνεια από τους Περουβιανούς και το σύστημά τους. Αλλά καταδικάζονται οι αδυναμίες του συστήματος που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Περουβιανοί το θέμα της χρηματοδότησης των ε, πολιτικών κομμάτων, που όπως είπε και ο Χαβιέρ Λόπες, το θέμα του εκλογικού νόμου, που είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα σύστημα ισχυρών κομμάτων, που σίγουρα είναι δυναμία της δημοκρατίας του Περού. Πάντως, ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, το ότι διαπιστώσαμε ότι η μεταρρύθμιση μπήκε και εισήχθη στη μέση της διαδικασίας, ε, κάτι το οποίο εμπόδισε κάποιους υποψηφίους να συμμετάσχουν στις εκλογές. Υπάρχει στη δήλωσή μας. Και όπως είπε και ο Λουίς Δεγκράντες, έτσι και εγώ πιστεύω ότι τα περουβιανά κόμματα και οι αρχές συνειδητοποιούν ότι χρειάζονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις, κάτι το οποίο ανοίγει το δρόμο σε σημαντική συνεργασία. Δεν είμαστε εμεί οι συντονιστέ βέβαια, εννοείται, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο μας να συνεργαστεί και να προτείνει σημεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να βελτιωθεί η δημοκρατία στο Περού. Κάτι το οποίο είπαμε και όταν ήμασταν εκεί. Τονίσαμε τις αδυναμίες δηλαδή του συστήματος η διαδικασία έχει αρχίσει. Από εκεί και πέρα και η τεχνική πτυχή της αντιπροσωπείας μας εκεί βοήθησε, τα επισήμανε όλα αυτά και θα προχωρήσουμε ανάλογα. Η κυρία Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δώσατε να πάμε ως παρατηρητές στην αντιπροσωπή αυτή και να έρθουμε εδώ να σας διηγηθούμε αυτά τα οποία είδαμε. Για μένα ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια τέτοια αποστολή. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Δεν είναι πάντα γνωστός, αλλά οι χώρες στις οποίες πάμε ως παρατηρητές είναι ευγνώμονες απέναντί μας για την παρουσία μας εκεί. Χαίρομαι λοιπόν που ο Αντιπρόεδρος Μπαλτάθερ θα αναλάβει στην κυβέρνηση Κοντίνσκι και θέλω να ευχαριστήσω τη Ρενάτε, την επακεφαλή στην αντιπροσωπεία μας για το έργο της, αλλά και όλη την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρουσία εκεί, αλλά και για το προπαρασκευαστικό έργο τους. Τώρα, η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι δεν μπορούμε να περιοριστούμε στην παρατήρηση των εκλογών. Τα αποτελέσματα του έργου μηνών περιλαμβάνει συστάσεις. Οι συστάσεις που υποβλήθηκαν λοιπόν μετά το δεύτερο γύρο των εκλογών, αλλά και μετά και από τον πρώτο, επιμένουν και υπογραμμίζουν το πρόβλημα που έχει το Περού, δηλαδή την αδυναμία των δημοκρατικών του θεσμών. Επειδή δεν είναι ισχυρά τα πολιτικά κόμματα, εξαιτία του συστήματος χρηματοδότησης, επιμένουν σε αυτό μάλιστα, και στο δεύτερο γύρο μιλήσαμε και για μεγαλύτερη κοινοβουλευτική συνεργασία. Ε, συμφωνώ, δεν ε, θέλουμε να δώσουμε μαθήματα σε κανέναν, αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε μια διαδικασία ε, τη στιγμή που και οι ίδιοι είπαν ότι θα θέλαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τους συνοδεύσει και να τους βοηθήσει στη διαδικασία. Αυτή λοιπόν είναι μια σκέψη πάνω στην οποία πρέπει να προβληματιστούμε. Και είναι σημαντικό γιατί ο πρόεδρος Κοτσίνσκι θα τα βρει πολύ δύσκολα τα πράγματα εξαιτίας αυτής της αδυναμίας πλειοψηφιών έχει τεράστιες προκλήσεις να αντιμετωπίσει η χώρα. Οπότε αφού αυτοί θέλουν τη συνεργασία και εμείς πρέπει να αναλάβουμε δράση και να φροντίσουμε να προσφέρουμε αυτή τη συνεργασία για να βελτιώσουν τη δημοκρατία τους και ώστε το Περού να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατότητα που έχει για να πάει προς τα μπρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Παντζέρη. Να ευχαριστήσω με την ε, σειρά μου την εισηγήτρια για αυτή την ε, εκλογική αποστολή παρατήρησης του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και θα μπορούμε να πούμε ότι οι εκλογές έγιναν με τρόπο συντεταγμένο, βιθαρχημένο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Θα πρέπει βέβαια να δούμε κάποια σημεία τα οποία προσέξαμε και επισημάθηκαν σήμερα. Είπαμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε κάποια θέματα στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο ήταν τα πράγματα απλούστερα από τον μόνο δύο υποψήφοι. Υπάρχουν κάποια θέματα λοιπόν που αφορούν τον εκλογικό νόμο. Ας πούμε στο Κούσκο είχαμε κάποιες άκυρες ψήφους και κάποια λευκά ψοδέλια δηλαδή που φτάνανε στο 35%. Εδώ και υπήρχε πρόβλημα πληροφόρησης. Επίσης θέλω να σταθώ και στην πρόσβαση των ΜΜΕ. Το δικαίωμά τους δεν ήταν τόσο προστατευμένο Υπήρχαν ε, κάποια όρια, αλλά τα όρια αυτά ε, για την περιφρούση των εκλογών σίγουρα παραβιάστηκαν. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπάψη, υπόψη ότι έχουμε διάφορους που ανακατεύθηκαν με τις εκλογές και προερχόντουσαν από τους κύκλους των εμπόρων ναρκωτικών. και πάρα πολλοί υποψήφοι κατέβηκαν στις εκλογές ως υποψήφοι για να αποφύγουν τη σύλληψη. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί βρισκόμαστε σε κάποια σίγουρα σπουδαία χώρα, αλλά υπάρχει πάρα πολύ εκτεταμένη παραοικονομία. Και γι' αυτό που είπε για τον ε, ε, και για το πώς έπιασε τόπο αυτή η ιδεολογία. Έπιασε τόπο γιατί ρίζωσε καλά στον χώρο της παραοικονομίας. Για να δούμε πάντως το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι μπορούμε να αισθανθούμε ανακούφιση. Κέρδισε βέβαια και ο Κατσίνσκι, αλλά και γιατί από τις ε, εκλογές φάνηκε ότι τελικά ο φουχημορισμός ήταν κάτι το αρνητικό και αυτό και βγήκε από το αποτέλεσμα που βγήκε στις φυλακές. Τώρα επομένως υπάρχει ένα καινούργιο όραμα για τη χώρα. Αυτό επίσης είναι άλλο δίδυμα της εκλογές. Ο όραμας μας ποιος είναι. Όχι μόνο το να βοηθήσουμε ε, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Ούτε πρέπει από καθέδρας να τους κουνάμε το δάχτυλο, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις οικονομικές, κοινωνικές και εκλογικές. Μόνο έτσι η χώρα θα μπορέσει να προοδεύσει πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που εγώ άντλησα από τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο από αυτήν την εκλογική μας εμπειρία. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Βέμπερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα σχόλια συγκλίνουν σε αυτή την ανάγκη να υπάρξει μια ευρεία και εδρεωμένη στην, ε, στο Περού, στο εκλογικό δίκαιο και σε άλλα θέματα και οι προτάσεις, οι συστάσεις μας της επόμενη εβδομάδα θα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η χώρα αυτή απαιτεί μεταρρυθμίσεις σε βάθος, όχι μονάχα σε εκλογικό επίπεδο, αλλά σε ό,τι αφορά το σύστημα των πολιτικών κομμάτων. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα, δεν υπάρχει κομματική ζωή εκεί. Σε κεντρικό επίπεδο ίσως, ελάχιστα, αλλά σε τοπικό επίπεδο είναι ολέθρια τα πράγματα. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Από τους 130, από τους 130 εκλεγμένους βουλευτές, 100 δεν ήταν μέλη των κομμάτων υπό την σημαία των οποίων κατέβηκαν. Αυτό είναι κάπως δύσκολο να το καταλάβει κανείς στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχει η έννοια της κομματικής πειθαρχίας, πώς θα ακολουθήσουμε τη γραμμή ενός κόμματος, ο έλεγχος που έχει ένα κόμμα στους βουλευτές του και πώς μπορεί να έχει έλεγχο πάνω σε αυτούς τους βουλευτές γιατί εμφανίζονται στις εκλογές, γιατί είναι, έχουν κάποια φήμη ή έχουν χρήματα ή οτιδήποτε τέτοιο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η μεταρρυθμίση σε επίπεδο εκλογικού δικαίου και νόμου των κομμάτων και εδώ το θέμα της χρηματοδότησης της πολιτικής ζωής στο Περού είναι κεφαλαιόδες γιατί είδαμε σε αυτές τις εκλογές πραγματική πολλές καταγγελίες ότι εμπλέκεται βρώμικο χρήμα, χρήμα από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών κτλ. Όταν έχει κανείς τέτοιες κατηγορίες, καταγγελίες, αυτό που είναι απαραίτητο είναι να εξασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια σε σχέση με τη χρηματοδότηση στις προεκλογικές εξαρτίες, είτε πρόκειται για κόμματα, είτε πρόκειται για ανεξάρτητους υποψηφίους και πρέπει να πω ότι κάπως οι πολιτικοί διστάζουν ή έχουν εμπόδια σε σχέση με τη διαφάνεια, σε σχέση με τη χρηματοδότηση που παίρνω από ιδιωτικούς φορείς. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να πιέσουμε για αυτό το θέμα. Να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν συμμαχίες με την κοινωνία των πολιτών, με τους δημοσιογράφους, με τα μέσα επικοινωνίας, ώστε να προωθήσουμε την ιδέα μιας μεταρρύθμισης στο Περού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τη χώρα αυτή. Και είμαι πεπισμένη ότι οι βουλευτές εκεί δεν θα δεχτούν μια εμβαλωματική θα, θα δεχτούν εν μια ε, τροποποίηση για να αποτραπεί αυτό το οποίο συνέβη στις τελευταίες εκλογές. Αλλά αυτό δεν είναι επαρκέ. Πρέπει να υπάρξει ευρύτερη μεταρρύθμιση. Χωρί μεταρρύθμιση στη χρηματοδότηση των κομμάτων δεν θα μπορέσουμε να βρούμε πραγματική πρόοδο στη χώρα αυτή. Και μακάρι όλοι να αποδεχθούν, θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα, μακάρι όλοι να δεχτούν αυτές τις ιδέες και πρέπει να το κάνουν το ταχύτερο δυνατό μέσα στο επόμενο εξάμεινο, πρέπει να εφαρμοστούν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα της τη διάταξης το οποίο είναι η έκθεση της κυρίας Φωτίγκα η νέα στρατηγική επικοινωνία για να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα που εκπορεύεται από τρίτες δυνάμεις. Η κυρία Φωτίγκα έχει το λόγο. Thank you, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη συζήτηση για την έκθεση αυτή. Μετά από πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε την πρώτη φορά που εξετάσαμε το σχέδιο αυτό ψηφίσματος. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα κρόαση που οργάνωσε η Επιτροπή μας, η ΑΦΕΤ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αρχίσω ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους Πρόεδρος, διακόπτη. Ησυχία παρακαλώ. Παρακαλώ κυρία Φαντίγκα. Έλεγα λοιπόν ότι θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους οι οποίοι συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην εκπόνηση του κειμένου αυτού. Πρόκειται για μια συνδυασμένη προσπάθεια, για μια συλλογική προσπάθεια που έκαναν μαζί οι σκιώδεις συζητητές με εμπειρογνώμονες από τη γραμματεία της ΑΦΕΤ, την κυρία Γιάννα Καμίνσκα για παράδειγμα. Θέλω να ευχαριστήσω και το δικό μου προσωπικό και τους συμβούλους του, της πολιτικής μου ομάδας για την ε, πολύτιμη συμβολή τους. 358 τροπολογίες υποβλήθηκαν στην έκθεση αυτή. Τρεις ε, φορές συνεδριάσαμε εξετάζοντας τις τροπολογίες προκειμένου να διαπραγματευτούμε συμβιβαστικές και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι το έργο αυτό απέδωσε. Καταφέραμε και συμφωνήσαμε επί 21 συμβιβαστικών τροπολογιών επί του κειμένου. δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Καταλήξαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, που πάντα είναι δύσκολο να βρει κανείς χρόνο εκεί. Κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν παραπάνω χρόνο για να εκτιμήσουν τις τροπολογίες και να συζητήσουν μεταξύ τους. Πάντως ευχαριστώ τη Γραμματεία που συμφώνησε τελικά. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω δύο σχόλια. Η συζήτηση κράτησε πολύ και μπορώ να πω ότι η συνεργασία μεταξύ μας οδήγησε στο τελικό κείμενο, αλλά μας βοήθησε προηγουμένως να δούμε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα που εξετάζουμε. Ένα ζήτημα κυρίως θα αναφέρω. Από την αρχή, δουλεύοντας για την έκθεση αυτή, θα έλεγα ότι βρεθήκαμε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέχρι και πίεση θα έλεγα από οργανώσεις μέσων ενημέρωσης ή ακόμα και λόμπις. Σπούτνικ και άλλοι έδωξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο δικό μας έργο. Από ολόκληρη την Ευρώπη θα έλεγα ενδιαφέρθηκαν για αυτό που κάναμε. Το πρακτορείο Σπούτνικ και τα λοιπά. Εμείς δεχτήκαμε από την αρχή, ήταν το μάντρα μας, ότι παρά τις όποιες προσδοκίες που περιλαμβάνονται στην στρατηγική μας για την ασφάλεια υπήρξαν απειλές και από την Ανατολή, ιδιαίτερα μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Ουκρανίας, λέει η ομιλήτρια, αλλά και στη Δύση, κυρίως με την άνοδο δύο ε, Ισλαμιστικών οργανώσεων, κυρίως της ΔΑΕΣ, του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις, ε, τις απειλές και από τις δύο αυτές πλευρές και μάλιστα συγχρόνως. Και να αναγνωρίσουμε ότι και οι δύο αυτές απειλές υπάρχουν παρόλο που είναι διαφορετικής φύσης και ο στόχος τους ίσως πάντως Στη μία περίπτωση πρόκειται για ένα κρατικό παράγοντα, στην άλλη περίπτωση πρόκειται για ένα μη κρατικό παράγοντα που χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία. Παρόλα αυτά, όσον αφορά την στρατηγική της επικοινωνίας μας, μπορούμε να εντοπίσουμε δραστηριότητες προπαγάνδας που έρχονται και από τις δύο πλευρές. Στην έκθεση αυτή λοιπόν γνωρίζοντας ότι πρέπει να αντισταθούμε στα επιχειρήματα της Ρωσίας, η οποία προσβλήθηκε που συνδυάσαμε τα δύο αυτά ζητήματα, τις δύο αυτές απειλές σε μία και την ίδια έκθεση. παρόλα αυτά πρέπει να δείξουμε ότι αντιστεκόμαστε σε αυτού του είδους την επιχειρηματολογία, δεν τη δεχόμαστε και να δείξουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα όλα τα προβλήματα, αναγνωρίζοντάς τα και βέβαια διαβλέποντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά στη μία και στην άλλη περίπτωση. Και θέλω αυτό να το πω στους συναδέρφους, γιατί κατά τη γνώμη μου τα καταφέραμε. Μετά από μακρές συζητήσεις, λαμβάνοντας υπόψη πολλά ιδιαίτερα περίπλοκα ζητήματα. Συνεπώς, ακόμα και κατά τη διάρκεια του έργου μας για την έκθεση αυτή, συνεχίσαμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις προκλήσεις, αλλά και να δρούμε με την πολιτική του μαστιγή και του καρότου. Πρώτα δεχτήκαμε την ανάγκη να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και να ψηφίσουμε από αυτού και να αξιολογήσουμε ε, τη δυνατότητα που έχουμε. Χτες είδαμε την ταινία αυτή της Λετωνίας. Είναι ένα ε, ντοκιματέρ στο Stratcom ε, από τη Βασοβία. Πρόκειται ε, μια προβολή που έκανε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βαρσοβία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον που δείχνει ομάδες, που δείχνει τις επιθέσεις, τα τρόλς επίσης. Χτες στο Russia Today μπόρεσα να δώσω μια συνέντευξη. Σπάνιο βέβαια, πολύ σπάνιο. Δεν θα ήθελα εγώ να χρησιμοποιήσω τέτοιου είδους καρότο. Η απειλή υπάρχει από το Stratcom και είναι μεγάλη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και σίγουρα μπορεί δυστυχώς να προσελκύσει την ολέα μας. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί ακόμα και νέα κορίτσια ε, μπορεί να προσελκυστούν και να προσχωρήσουν σε τέτοιες Ισλαμικές οργανώσεις. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τα μέσα, να δείξουμε την ε, αντοχή μας και τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Γι' αυτό ζητώ από τους συναδέρφους να συνεχίσουν το έργο και να στηρίξουν την έκθεση αυτή. Να συνεχίσουμε με το ίδιο θετικό πνεύμα και ευχαριστώ και πάλι όλους τους σκιώδες εισηγητές χωρίς καμία εξαίρεση. Η συνεργασία ήταν εξαιρετική. Πολύ μου άρεσε που μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί σας. Μία από τις πολιτικές ομάδες μου είπαν ότι θα ήθελε να παρουσιάσει τη δικιά της έκθεση μειοψηφία. Που σημαίνει ότι στη συμβαστική, στο συμβαστικό κείμενο δεν αντικατοπτρίζεται η δικιά τους άποψη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους κοιοδησηγητές, πρώτα τον κύριο Ουγγουράνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να συμφωνήσω μαζί της αυτή η έκθεση δεν είναι μια μορφή εξίσωσης της Ρωσίας με τον ΤΑΕΣ, το ΆΕΣΙΣ. Είναι μια έκθεση που αφορά την προπαγάνδα. Θα έλεγα μία προπαγάνδα και δύο προπαγανδιστές. Επομένως αφορά και τις δύο αυτές δυνάμεις, τη Ρωσία και το Ισλαμικό κράτος. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά στις συναντήσεις των σκιωδών και νομίζω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή. Ξέρω ποια είναι τα προβλήματα της προπαγάνδας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι μια πολύπλοκη μορφή προπαγάνδας. Κατανοώ γιατί οι πολιτικές ομάδες χρειάστηκαν χρόνο για να συγκεντρωθούν σε αυτό το πρόβλημα. Πάνω απ' όλα όμως μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι μια έκθεση που αφορά την αντιευρωπαϊκή προπαγάνδα είναι πια μια πραγματικότητα η Ευρώπη αντιμετωπίζει πράγματι α, παραπληροφόρηση σε τεράστια κλίμακα από τόσο, τόσο από και μη κρατικούς φορείς. Και ελπίζω ότι μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές θα βρούμε κοινό έδαφος. Θα έχουμε περαιτέρω συναντήσεις για να οριστικοποιήσουμε αυτή την έκθεση Αυτή η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ψηφίσει πολλές εκθέσει όπου αναφέρονται τα θέματα της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Μια πλήρη έκθεση για τον αγώνα κατά της προπαγάνδας είναι το επόμενο λογικό βήμα. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Προεδρεύων. Ο Φρόντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Μιχαήλ. πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για μένα να βρεθώ σαν σκιώδης εισηγητής αντιμετωπίζοντας ένα τόσο, μια τόσο ισχυρή προσωπικότητα την Μάργαρετ Θάτσερ ή αλλιώς γνωστή ως ε, Αναφωτίγκα ως αντίπαλο. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζει κανείς την κυρία Φωτίγκα. Νομίζω ότι καταφέραμε να συνεργαστούμε όμως όσο καλύτερα μπορούσαμε και θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Τούτου λεχθέντος βέβαια, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια θέματα όπου δεν μπορέσαμε να βρούμε πλήρη σύμπνοια πρώτα απ' όλα. Και αυτό είναι το θέμα με το οποίο έχω κάποιο πρόβλημα. Είναι ο συνδυασμός της προπαγάνδας της Ρωσίας και του Ισλαμικού κράτους σε μία έκθεση. Γιατί, το είπα αυτό και από την αρχή, γιατί αυτό το οποίο θα κάναμε, συνδέσουμε, συνδυάσουμε αυτές τις δύο πτυχέ και δεν το έχουμε κάνει ακόμα γιατί δεν έχουμε δημοσιεύσει αυτή την έκθεση ακόμα, ουσιαστικά θα ανυψώσουμε το Ισλαμικό κράτος στο ίδιο επίπεδο όπως και η Ρωσία. Κάτι λοιπόν το οποίο θέλουμε να αποτρέψουμε και είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αναγνωριστεί το Ισλαμικό κράτος ως κράτος ή ως ιονή κράτος, βλέπω να είστε κοινών το κεφάλι σας κύριε Φωτίγκα. Αλλά και πάλι δεν βλέπω πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα αλλιώς. Προς το όφελος της ε, συνένωσης των επιχειρημάτων μας. Κάποια ακόμα πράγματα. Για μένα είναι σημαντικό. Να έχουμε ένα σωστό ορισμό της προπαγάνδας, να ορίσουμε τι σημαίνει προπαγάνδα, ώστε να είναι σαφές για όλους μας τι ακριβώς εννοούμε. Θα πρέπει να κατανοήσουμε επιπλέον ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά συναισθήματα σε σχέση με το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει αυτή η προπαγάνδα επί των πολιτών των κρατών μελών. Πρέπει επίσης να κάνουμε και διάκριση μεταξύ της κακής προπαγάνδας και της καλής πληροφόρησης. Θα πρέπει να διακριβώσουμε ακριβώς πώς επηρεάζονται οι πολίτες μας από αυτό το είδος προπαγάνδας. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο πρακτορείο Σπούτνικ, το οποίο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στην παρουσίαση αυτής της ταινίας που προβλήθηκε χθες. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο το έργο αυτό ή γενικά οι διαβουλεύσεις μας για τα θέματα αυτά. Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτό σε τι οδήγησε. Εσείς μπορείτε να δείτε, να το γράφει αυτό το Sputnik, γιατί <clears throat> παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του. Αλλά μπορεί οι υπόλοιποι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν πάρει πρέφα. Δεν διαμφισβητώ το γεγονό ότι έχετε κάθε λόγο να είσαστε ενδιαφερόμενοι για τα θέματα αυτά. Τελικά ποιο νοιάζεται για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν λέω ότι κανεί δεν ασχολείται με το θέμα αυτό. Απλώ δεν ξέρουμε ποιο παρακολουθεί αυτά τα πρακτορία, αυτέ τι ιστοσελίδε. Δεν ξέρουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η προπαγάνδα, γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια δημοσκόπηση ή κάποια έρευνα, κάποια προσπάθεια να κάνουμε μια μελέτη του αποτελέσματος αυτού. Αν δούμε ότι υπάρχουν 10 εκατομμύρια Πολωνοί που βλέπουν κάθε μέρα το Sputnik, κάθε μέρα δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα ήθελα όμως να ξέρω <clears throat> πρωτού προχωρήσουμε σε αυτή τη διατύπωση. Και εν τέλει θα ήθελα να σας ζητήσω το εξή <clears throat> γιατί είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και υποτίθεται ότι θα πρέπει να διεκπεράσουμε αυτό το θέμα την πρώτη μέρα ουσιαστικά μετά από τις διακοπές. Και έχουμε ακόμα μεγάλες αποστάσεις σε σχέση με πολλά από τα θέματα. Θα ήθελα να σας ζητήσω μήπως <clears throat> μπορούμε να καθυστερήσουμε το θέμα αυτό ώστε να το αντιμετωπίσουμε λίγο αργότερα την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές γιατί από σήμερα μέχρι τις 29 Αυγούστου δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν λίγο περισσότερο χρόνο για να σκεφτούμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Αυστρεβίτσιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι με μεγάλη ικανοποίηση μελέτησα όλα όσοι έχουν σχέση με το θέμα μας. Είναι μεγάλη πρόκληση και είναι νοπές ακόμα οι εντυπώσεις γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ενεργειακής ασφάλισης αλλά και της κυβερνοασφάλειας. Κανείς πλέον δεν αμφισβητεί αυτές τις έννοιες. Αλλά πολλοί εξημών δεν πιστεύουν ότι η ασφάλεια για την πληροφορία και ενημέρωση ή ε, της ανεξάρτητης των πληροφοριών είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την ασφάλεια. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να ευχαριστήσω για αυτήν την έκθεση ιδίας που ήρθε την κατάλληλη ώρα, που αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε και να συζητούμε, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, αλλά τελικά ετέθηκε της τραπέζης το εν λόγω θέμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης, κανείς λόγος να αγνοούμε την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα. Πρόκειται για μια πρόκληση που έχει επιτεθεί, έχει, έχει θίξει τις δυτικές αξίες. Και είναι κάτι πάρα πολύ δυσάστατο το οποίο συμβαίνει ολόγυρα. Όντως η προπαγάνδα είναι μη δημοκρατικό μέσο, κατασταλτικό, καταπιεστικό και αυταρχικό. Το χρησιμοποιούν και οι, οι τρομοκρατικές οργανώσεις για να προβληθούν προς το κοινό και έχουμε επίσης κάποια κρατικά μέσα ενημέρωσης τα οποία ξέχασαν για ε, τα κράτη τους ξέχασαν τι θα πει το κρατικό ραδιόφωνο και η κρατική τηλεόραση γιατί εδώ στη γειτονιά μας έχουμε κάποιες χώρες που νομοθετικά αλλά και de facto ε, τέτοια μνημιέ κρατικά είναι η πραγματικότητα. Επομένως δεν μπορεί κανένας να έχει κάποια ένσταση ότι έχουμε κάποια, ε, κάποιο κρατικό κανάλι το οποίο το ελέγχουν ε, οι αρχές της χώρας και όποιος γενικά έχει το συμφέρον του να επίτηδες να διαδίδεται κάποια συγκεκριμένη προπαγάνδα. Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση και όχι πληροφόρηση. Ποιος το αμφισβητήσει αυτό. Δεν βλέπω συνάδελφοι καμία διαφορά μεταξύ των εμπλεκόμενων στο, στα ΜΜΕ κατά αυτόν τον τρόπο που είναι το κράτος ε, ή όταν δεν είναι το κράτος. Γιατί τελικά ε, το θέμα κλειδί είναι τα χρηματοοικονομικά. Και έχουμε κάποια κράτη που το κάνουν αυτό, έχουμε κάποιες τρομακτικές οργανώσεις που είναι σε διάφορες ε, περιοχές και που σαν τμήμα του υβριδικού πολέμου που κάνουν ασχολούνται και με την προπαγάνδα. Τελικά είναι κάτι σαν ορολογιακή βόμβα γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα εκραγεί. Έτσι κανείς μπαίνει στα μυαλά των ανθρώπων, τους κάνει πλήση εγκεφάλου και στη συνέχεια έχει έφορο έδαφος για λάθος αντιλήψεις και λάθος αποφάσεις. Όλοι μας καταναλώνουμε την πληροφορία. Ίσως δεν υπάρχει κανείς πάνω στη γη που δεν ε, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Οπότε γι' αυτό και η προπαγάνδα ενεργεί με αυτόν τον τρόπο και έχει τόσο σημαντικές επιπτώσεις ε, πάνω στους ανθρώπους και σας το λέω ξεκάθαρα. Ε, τι θα γίνει, θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση επίτροπο προπαγάνδας ή κάποια άλλη πλατφόρμα, κάποιο, κάποια υπηρεσία. Όχι, αυτό το απορρίψαμε θέση εξ αρχής γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να είναι μη αυτοεκπληρούμενη η προφητεία και γι' αυτό και δουλέψαμε σκληρά για να βρούμε κάποιες συμβαστικές λύσεις. Να, και το κείμενο αυτό ίσως ε, θα πρέπει να αλλιώ για την ψηφοφορία. Ίσως οι διορθωτές του κειμένου, οι αναθεωρητές του κειμένου, ίσως το ε, έκαναν συντομότερο, υπήρχαν κάποια θέματα εκεί. Αλλά νομίζω ότι η ουσία του κειμένου είναι αρκετά αξιόλογητος ώστε να είναι βάση για προβληματισμό. Επίσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο ε, την ανεξάρτητη δημοκρατία στην Ευρώπη γενικότερα και ειδικότερα ε, στην ε, γειτονιά μας, γιατί εκεί στηρίζονται οι αξίες της Ευρώπης. Αυτορύθμιση, αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε έναν big brother, έναν μεγάλο αδερφό που να τι θα σέβει τα ΜΜΕ. Γι' αυτό και κατέληξαμε σε αυτή την πρόταση να υπάρξει δηλαδή κάποιο είδου οδηγία της Ένωσης. Θα πρέπει να γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις γιατί δεν χρειαζόμαστε ιδεολογικά μέσα, χρειαζόμαστε νομοθετικά μέσα για να κατοχυρώσουμε μια πληροφορία και πληροφόρηση αντικειμενική, ελεύθερη, συγκρίσιμη. Στην συνάντηση κορυφή της ε, Βαρσοβίας που μόλις ολοκληρώθηκε, πρόκειψε στενότερη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων που ασχολούνται με την ασφάλεια στην κοινωνία που ζούμε. Γι' αυτό και είναι κάτι αξιόλογο το κέντρο αριστείας που τώρα θα εδρεύει στην ε, Λετωνία και η Stratcom επίσης είναι πολύτιμη γιατί αποτελεί κάποια μικρή ομάδα που έχει εμπειρογνωμοσύνη και μπορούν εκείνοι να αναγνωρίσουν μέσα άσκησης προπαγάνδας τα οποία ε, μας τα έχουν πετάξει και εξαπολύσει εναντίον μας. Ξέρω δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους, τη Γέση Χάρο, η οποία εργάζεται για το Ούλε, ένα κανάλι της Φιλανδίας και την ε, Άντεν που προέρχεται από την Γερμανία. Οι δύο είναι υπέροχες, εγωιτευτικές και επαγγελματίες δημοσιογράφοι, οι οποίες κατέγραψαν το πώς τους ε, έριξαν τρολάρισμα, πώς τις ε, εκφόβησαν, χειρότεροι ε, συνανθρωποί μας. Όμως, αυτά τα οποία είπαν αυτές οι δύο δημοσιογράφοι, μόνο κάποιοι που είναι τυφλοί και κουφοί δεν μπορούν να τα προσέξουν και να τα ακούσουν. Γιατί ακριβώς όσο περισσότερο αρνούμεθα και δεν διακρίνουμε αυτήν την εχθρική προπαγάνδα που κατευθύνεται στη δυτική μας κοινωνία, τότε τόσο περισσότερο θα κινδυνεύουμε γιατί θα πρέπει να αντιδρούμε σε αυτήν την προπαγάνδα, συνάδελφοι. Απόψε θα έχουμε μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα γίνει προβολή κάποια ταινίε για την υπόθεση Μαγνίτσκι. Πρόκειται για μια προσπάθεια παραπάνω που αφορά την απόπειρα αμάβρωσης της μνήμης του Μαγνίτσκι. Πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια προπαγάνδας και προπληροφόρησης. Αυτοί που έφτιαξαν αυτή την ταινία έχουν τους λόγους τους, έχουν τους σκοπούς τους. Να μαυρώσουν την φήμη του προσώπου αυτού, να μας κάνουν να τον αγνοούμε. Θα πρέπει να πούμε όχι στην προπαγάνδα. Οπότε ας το δούμε έτσι, έτσι όπως μας το σερβίρουν. Άρα σίγουρα δεν είμαστε στο πλευρό τους και πάλι ευχαριστίες θερμές στην Άννα για την πρωτοβουλία της. Ο Γκάλιας, δίνω ρόλο στην κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Φωτίγκα, διότι όλοι καταλαβαίνουν. Πρόκειται για τη δημοκρατία στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς πάντα είμαστε υπέρ του πλουραλισμού και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, αλλά δεν είναι εύκολο να συζητάμε ε, τέτοια ζητήματα όταν υπάρχει πολύ καλά οργανωμένη προπαγάνδα σε μία ή την άλλη γείτονα χώρα μας. Δεν έχει νόημα να αρνηθούμε ότι η Ρωσία κάνει οργανωμένη επίθεση προπαγάνδας σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης. Μια λοιπόν από τις βασικές ιδέες της συζήτηση για την ομάδα μου αλλά και για άλλους συναδέρφους είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την ισορροπία που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε από τη μια την ελευθερία τύπου και το πλουραλισμό αλλά από την άλλη να προστατεύσουμε και τα συμφέροντά μας σε αυτού του νέου είδους αναπτυσσόμενη αντιπαράθεση μέσω της προπαγάνδας. Στον κύριο Φρόιντ θέλω να πω κάτι πριν περάσω στις λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι είναι όλα όπως τα λέτε. Δεν βάζουμε στο ίδιο επίπεδο το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος με τη Ρωσία. Κανένας δεν βλέπει το Ισλαμικό κράτος σαν του ίδιου είδους οργάνωση όπως είναι το κράτος της Ρωσίας. Η... Το μοντέλο όμως μάλλον και τα μέσα που χρησιμοποιούνται ψηφιακά μέσα ενημέρωσης που είναι στη διάθεση όλων τελικά τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι παρόμοια και το μοντέλο που χρησιμοποιούν η μία και η άλλη πλευρά είναι παρόμοια. Το συζητήσαμε ξανά και ξανά πώς να αντιμετωπίσουμε δύο διαφορετικούς φορείς, παράγοντες μάλλον, στον τομέα της προπαγάνδας. Δεν νομίζω ότι τους θεωρούμε ίδιους. Ούτε κανένας μεταξύ των σχεδόν, η συγγήτρια, δεν θέλησε να βάλει το κράτος της Ρωσίας στο ίδιο επίπεδο όπως το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, το Ντάσο. Ίσως θα έπρεπε προσεκτικά να το συζητήσουμε γιατί ίσως υπάρχει κάποια παρεξήγηση εδώ. Πάντως, πρώτον, είναι πολύ σημαντικό με την έκθεσή μας να στηρίξουμε τη δημιουργία μιας Γενικής Διεύθυνσης Stratcom. Ήταν καλή απόφαση αυτό. Συγχρόνως, αυτό το μικρό τμήμα υπό την κυρία Μογκερίνη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πραγματικά τα προβλήματα που διαπιστώνουμε. Πέρα από αυτά που συζητάμε υπάρχει μία διαδικασία για να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα ποιος τελικά θα είναι ο στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Stratcom και τι θα πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο χωρών μελών. Πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε τις δυνατότητες που διαθέτουμε να ενισχύσουμε τις κοινωνίες μας ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα την απειλή αυτή της παραπληροφόρησης. Γιατί στην στρατηγική προπαγάνδας το πιο πετυχημένο είναι η διάδοση της παραπληροφόρησης. Είτε δημιουργώντας συμμάχους, είτε δημιουργώντας αβεβαιότητα, είτε απλώς διαδίδοντας ε, ψεύτικες διαβεβαιώσεις. Οπότε πώς να διαχωρίσουμε την πληροφόρηση και την ελευθερία έκφρασης από την συστηματική παραπληροφόρηση και κυρίως στα πλαίσια της Ρωσίας που οργανώνεται από αυτούς που εργάζονται για τη Ρωσία, είτε με το Russia Today ή με το πρακτορείο Sputnik. Όποτε η ερώτηση είναι, ό,τι και αν πιστεύετε για την προπαγάνδα, στη Ρωσία, άπαξ και ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος με τις πολιτικές αποφάσεις στη Μόσχα. Εσείς τι νομίζετε ότι θα συνέβαινε αν κάποιο γερμανικό πρακτορείο πήγαινε εκεί και πρόσφερε δουλειά σε 40 δημοσιογράφους για να καταπολεμήσουν τα όσα λέει η Μόσχα. Αυτό πώς θα σας φαινόταν. Θα ήταν εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο στη Ρωσία. Λοιπόν, εμείς είμαστε ανοιχτοί και είναι καλό το ότι η Ευρώπη είναι ανοιχτή. Είμαστε πολύ ανοιχτή και στις δραστηριότητες των ε, μέσων ενημέρωσης. Το άκουσα σήμερα, δεν ξέρω αν πρόκειται για διαδόσεις, αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά άκουσα σήμερα ότι το Sputnik προσφέρει νέες θέσεις για 40 δημοσιογράφους στο Διβούργο. Αν αυτό ισχύει, είμαι πεπισμένη ότι γνωρίζω γιατί το κάνουν μπορεί να χρειάζεται για περισσότερη ελευθερία τύπου στη Σκοτία, μετά μάλιστα την απόφαση του Brexit. Μπορεί να μην υπάρχει στη Σκοτία αρκετή ελευθερία τύπου, δεν ξέρω. Αλλά γιατί το κάνουνε. Γιατί βάζουν τόσα πολλά χρήματα, γιατί θέλουν να πληρώσουν δημοσιογράφους για να δουλεύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε τα προγράμματα, τα ρωσικά και στο εξωτερικό των Ρώσων, θα δείτε τις διαφορές που υπάρχουν. Συνεπώς, το συμπέρασμα της συζήτησης για το ζήτημα αυτό είναι ότι ποτέ δεν θα δεχτούμε να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα με προπαγάνδα. Όμως, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πάρουν στα σοβαρά την κατάσταση. Να ενισχύσουν τις κοινωνίες μας, να ενισχύσουν τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και να παρατηρήσουν πολύ καλά το τι συμβαίνει. Δεν είμαστε στο τέλος αυτής της συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα ζητήματα που προέκυψαν στους σκιώδεις εισηγητές διαπιστώνουμε ότι είμαστε στην αρχή μόνο της διαδικασίας και θα δούμε και άλλες εκθέσεις και άλλες συζητήσεις με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριο να έχει το λόγο. Ευχαριστώ Μάρκελ που μου δίνετε το λόγο. η αντιμετώπιση της κυρίας για να συμπεριλάβει δηλαδή όλες τις πηγές ε, απειλής σε επίπεδο πληροφόρησης είναι κάτι το οποίο μπορώ να το χαιρετήσω και τη Ρωσία από την μια και τις ακεραιόφρονες Ισλαμικές δυνάμεις από την άλλη πλευρά, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ δύο αυτών των κινδύνων, των δύο αυτών κινδύνων καλύτερα. όταν πρόκειται για τον πόλεμο της πληροφορίας το Ισλαμικό κράτος και προηγουμένως η Ταλιμπάν και άλλες Ισλαμικές δυνάμεις είχαν βασιστεί πολύ λιγότερο στην πληροφορία από τη Ρωσική Ομοσπονδία και για ένα πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Αν πάρτε τον πόλεμο πληροφορίας που διεξάγει η Ρωσία οι πληροφορίες αυτές κατευθύνονται στην Ευρώπη. Και αυτό γίνεται εδώ και 100 χρόνια, του χρόνου θα είναι 100 χρόνια. Από την Μεγάλη Οκτώβριανή Επανάσταση στη Ρωσία. Και η επανάσταση αυτή ξεκίνησε το κύμα από πληροφόρησης που συνεχίστηκε επί 100 χρόνια. Θυμηθείτε το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Θυμηθείτε το πόλεμο στην Τσετσενία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαμε μεγάλες προσπάθειες παραπληροφόρησης από την ρωσική πλευρά. Ποιοι το κάνουν αυτό. Το κάνουν αυτοί που έχουν στη διάθεσή τους εξελιγμένους, εξελιγμένες μεθόδους που η Ρωσία τις έχει χρησιμοποιήσει σε πολύ ψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια με την KGB και άλλους φορείς είναι το μακρύ χέρι της ΚΑΓΕΜΠΕ. Υπάρχει η ίδια έδρα, η φυλακή της Λουμπλιάνκα στην Μόσχα. Εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους. Παραπληροφόρηση, η ψευδολογία είναι τμήμα της επίσημης ρωσικής πολιτικής χωρίς κανένα όνειδος. Ακόμα και οι υψηλότεροι αξιωματούχοι στην Ρωσία είναι χωρίς ντροπή. Ε, επομένως αυτή η έκθεση θα πρέπει να υπογραμμίσει ότι ο κίνδυνος αυτός για την παραπληροφόρηση είναι πολύ πιο σημαντικός από την πλευρά της Ρωσίας από ότι από την πλευρά του Ισλαμικού κράτους. Το Ισλαμικό κράτος έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Μας απειλούν με ένα φρικτό και βίαιο πόλεμο. Μας απειλούν να φέρουν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες στην Ευρώπη και να θέσουν σε κίνδυνο τη συνοχή της Ευρώπης. Αλλά ο μάστορας στην παραπληροφόρηση είναι η Ρωσία και έχει σταθεί ο ηγέτης στον τομέα αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Και από αυτή την πλευρά θέλω να αναφερθώ στη συμβαστική τροπολογία 16. Ο κύριος ε, Πόρτμαν συζήτησε μαζί μας πρόσφατα και συζητήσαμε για την χρηματοδότηση αυτών των ενεργειών που τροφοδοτούν τη ρωσική προπαγάνδα και μας είπε δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα τη ρωσική προπαγάνδα έχουν ε, χιλιάδες δολάρια στη διάθεσή τους και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Γι' αυτό στην τροπολογία 16, συμβαστική τροπολογία 16 και το χαιρετίζω, αναφέρουμε την ανάγκη να δημιουργηθεί μια χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού η οποία θα μας δώσει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την ρωσική προπαγάνδα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα αντιμετώπιση αυτής της προπαγάνδας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο, ο πρόεδρος. Κύριε Γιούρεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ είμαι, πεπισμένος, βαθιά πεπισμένος ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Η έκθεση αυτή δεν πρέπει να εξυπηρετήσει την προάσπιση των συμφερόντων μας και της ασφάλειές μας, αλλά είναι και πολύ σημαντική για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ θέλω να σταθώ σε αυτά τα οποία λέγονται στην δέκατη συμβιβαστική τροπολογία. Μετά το κομμουνιστικό μετά την κομμουνιστική εποχή έχουμε δύο δομές οι οποίες δημιουργήθηκαν αν διαφορετικές. Έχουμε καταρχήν την, ε, τους κάτοχους εξουσίας που έχουν μεταμορφωθεί σε μια ελίτ και αυτή η ελίτ έχει αποκομίσει το μονοπόλιο της εξουσίας στη Ρωσία. Και επίσης έχουμε τους πολίτες που είναι κατά κάποιο τρόπο ξεριζωμένοι, δεν καταλαβαίνουν πια τι γίνεται στη χώρα τους, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται σε διεθνώς επίπεδο, δεν μπορούν να καταλάβουν το καλό από το κακό. Γι' αυτό η Ρωσία χρησιμοποιεί την προπαγάνδα για να μιλήσει για την επιθετική δύση. Αυτή είναι η μυθολογία με την οποία τροφοδοτεί τους πολίτες ότι η Δύση θέλει να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη σε βάρος της Ρωσίας. Στην τροπολογία 10 λοιπόν υπενθυμίσουμε ότι αυτή η διαδικασία της κατά κάποιο τρόπο πολιτισδυτικής εκρίζωσης θέλουν να κάνουν τους ανθρώπους να ξεχάσουν τις πολιτιστικές τους ρίζες για να γίνουν πιο ευάλωτοι στην προπαγάνδα τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνδυάσουμε αυτή την τροπολογία με τις τροπολογίες του κ. Κόβατσεφ όπου αναφέρονται συγκεκριμένες αιτήσει ώστε να διατηρηθεί η μνήμη των εγκλημάτων της κομμουνιστικής περίοδου. Γιατί αυτό είναι και ένας φραγμός που μας που εμποδίζει την προπαγάνδα, που αναχαιτίζει την ρωσική προπαγάνδα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη και ένα ακόμα βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η ελίτ της ε, σημερινής Ρωσίας προήλθαν από την Σοβιετική Ένωση και επομένως η πολιτική τους εδράζεται στο ότι υπόσχονται στον πληθυσμό θα ξαναγίνει η Ρωσία μια μεγάλη δύναμη και στο μέλλον. Αυτός ο φόβος λοιπόν για να καταγγείλουμε τη ρωσική προπαγάνδα δεν πρέπει να συνεχιστεί μεταξύ μας. Θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν μια επιθετική δύναμη προκάλεσε πολέμους, εισέβαλε σε άλλες περιοχές στην Ευρώπη και επί 50 χρόνια κράτησε το μισό των κρατών μελών μας όμοιρους και δεν τους επέτρεψε να εργαστούν και να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους μας. Μιλάμε πολύ για την Ρωσία, αλλά δυστυχώς δεν μιλάμε για τη Σοβιετική Ένωση. Πρέπει λοιπόν να προσθεθούν όλα αυτά και νομίζω με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί πολύ καλή έκθεση τη κυρία Φωτίγκα. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρε, Εγώ ο κύριο Φρόιντ. Τελευταίο ομιλητή είναι ο κύριο Βάιγκλ. Σα ευχαριστώ. Ε, έχουμε αυτό το θέμα το οποίο είναι λεπτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή. Γιατί αυτό το θέμα <clears throat> έχει επίπτωση στην έννοια της πληροφόρησης ευρία τη έννοια. υπάρχει παραπληροφόρηση που μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Και αυτό πρέπει να είναι μια πτυχή της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προάσπισης των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Γι' αυτό πιστεύω ότι η βασική αντίληψη που διατρέχει αυτό το έγγραφο δεν είναι ορθή για ένα απλό λόγο. Υπάρχει, υπάρχουν πολλοί συναισθηματικοί λόγοι για να αντιμετωπίσει κανείς την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε διαφορετικές ίσως απόψεις για την εκτίμηση της κατάστασης στην Ευρώπη και στον περιγυρό της. Και αυτά δεν μπορούν να τεθούν στο ίδιο επίπεδο με την απειλή του Ισλαμικού κράτους. έχουμε πολλές παρεξηγήσεις και λαθασμένε αντιλήψεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και πρέπει εμείς να μπορέσουμε να ξαναβρούμε ένα σωστό έδαφος για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλαμικό κράτος. Ο παραλληλισμός μεταξύ Ρωσίας και ΝΤΑΕΣ νομίζω ότι δεν είναι ικανοποιητικός. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να, να σκεφτούμε για θέματα αυτής της έκθεσης και να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο χρόνο ώστε να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της τεχνολογίας, της πληροφόρησης και της στρατηγικής πληροφόρησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αντιταχθούμε στις προπαγανδιστικές επιθέσεις που χρησιμοποιούν τρομοκρατικές οργανώσεις γιατί χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτές οι οργανώσεις και είναι ιδιαίτερα επιδέξεις στο θέμα αυτό. Ενώ οι χώρες της Δύσης δεν έχουν αντίστοιχο μηχανισμό. Είναι λοιπόν στο χέρι μας να αποκλείσουμε όλες αυτές τις επιθέσεις προπαγάνδας από τον δικό μας χώρο και επίσης να δώσουμε την πραγματική εικόνα της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έκανε λοιπόν το UKIP στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατάφερε με ψευδείς πληροφορίες να οδηγήσει τους Βρετανούς σε μια πλειοψηφία η οποία υπεστήριξε το Brexit πολλοί από τους, μεγάλους, από τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανής τώρα έχουν μετανιώσει για αυτή την απόφαση που πήραν για το Brexit όταν αυτή η πληροφορία βασίστηκε σε λαθασμέ... αυτή η απόφαση βασίστηκε σε πληροφορίες με τις οποίες βομβαρδίστηκαν. Δεν θέλουμε λοιπόν να ε, δούμε να γίνεται κάτι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλοί πολίτες επίσης στη Μεγάλη Βρετανία που είχαν μια λαθασμένη εικόνα σε σχέση με τον πόλεμο του Ιράν και πάλι λόγω προπαγάνδας. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τις χώρες μας από συστηματική χειραγώγηση μέσω της προπαγάνδας. Αλλά υπάρχουν πολλές πληροφορίες οι οποίες διαδίδονται και γι' αυτό θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις πηγές πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να προτείνω να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το θέμα των πολλών πληροφοριών που έρχονται από την Ρωσία. Και πιστεύω ότι υπάρχουν ε, λόγοι να έχουμε μια πιο στεναρή αντιμετώπιση στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τη ρωσική προπαγάνδα. Εγώ βλέπω μερικές φορές το, το κανάλι Russia Today <clears throat> και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι ένα εργαλείο χειραγώγησης. Και εγώ θα το γνωρίζω αυτό και γι' αυτό γελώ με την αφέλεια αυτής της προσπάθειας χειραγώγησης η οποία γίνεται. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση Άρα, ποια είναι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια στον κόσμο εδώ στις χώρες μας. Θα πρέπει επομένω να τα πούμε έξω από τα δοντία. Να μην ρίχνουμε το φταίξιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουν οι εθνικέ κυβερνήσει, κατηγορούν τι Βρυξέλλε. Και εμεί ίδιοι τα κάνουμε αυτά. Τώρα. Σήμερα κιόλας πήγα σε κάποια συνάντηση. Και εκεί τι λέγανε. Ότι οι Ευρωπαίοι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να σταματήσουν να βρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι διεφθαρμένη. Μα εμείς θα πρέπει να σταματήσουμε να δικαιολογούμε κάποιες χώρες που εξαπολύουν προπαγάνδα και έχουν πρόβλημα διότι καταπατούν την ελευθερία της έκφρασης, καταργούν την ελευθερία του τύπου και κατανοώ ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ευαισθησίες που δεν υπάρχουν στην Ρωσία. Ε, πολλές φορές επίσης δείχνουμε ιδιαίτερη υπομονή και ανοχή, αλλά να βάλουμε πρώτα το συμφέρον μας και το συμφέρον του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Βάγγελ. Όπως ξέρετε δεν μπορώ να είμαι αμερόληπτο για αυτό το θέμα. Πρέπει βέβαια να είμαι αμερόληπτο μια που προεδρεύω. Τέλος πάντων θα πρέπει τώρα να ζητήσω από την κυρία Φωτίγκα να δευτερολογήσει αλλά να μην πάρει περισσότερο από λίγα λεπτά γιατί έχουμε και άλλο θέμα στη μέρη διάταξη. Φωτίγκα, Σα ευχαριστώ. Σίγουρα και πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν μέρος σε αυτή την συναρπαστική συζήτηση και μας είπαν τι τους απασχολεί και πώς το σκέφτονται. Είδαμε από την συζήτηση ότι πραγματικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που είναι πολύ περίπλοκο. Πρόκειται για μεγάλη απειλή, πρόκειται για απαράδειτες συμπεριφορές. Πρόκειται επίσης και για ε, πηγή του προβλήματος που είναι μη κρατικότητος όπως ε, ε, το ΝΤΑΕΣ. Από την άλλη μεριά έχουμε και τέτοια δραστηριότητα παραπληροφόρησης και από κράτη ε, η δράση τους αυτή οδηγεί σε αποσταθεροποιητική ενημέρωση και σε κάποιο στραβλή εντύπωση που αποκομίζουμε στη καθημερινή μας ζωή. Και ξέρετε, ακόμα και κατά αυτή την περίοδο που δούλευα για αυτό το κείμενο, διαπίστωνα πώς οι Ρώσοι προσπαθούσαν να λιώσουν την ενημέρωση ακόμα και μέσα από αξιοσέβαστα ΜΜΕ. Προσπαθούσαν να επηρεάσουν τα πράγματα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Κύριε Φρόιντ, μας μιλήσατε για το Σπούτνικ κατόπιν των όσων σας είπα εγώ και αμφισβητήσατε την ε, επιρροή που ασκεί λόγω του, του, περιορισμένου βεληνικούς που έχει. Δεν ε, ε, δουλεύουν στην Πολωνία, αλλά αλλού. Ας πούμε στην ε, Αυστρία. Και ακριβώς όχι επειδή έχει τόσο μεγαλοβεληνικές, αλλά πάντως είχαμε και την Στράτκο ε, που επίσης ήταν πάρα πολύ επιδραστική και στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και έτσι προέκυπταν ε, ενημερωτικά δελτία που τα παίρνανε άλλα ΜΜΕ, οπότε έτσι υπήρχε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Άρα αυτό το οποίο επιβάλλεται είναι να υπάρξει ποιοτική δημοσιογραφία. Πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε τελικά να υπάρξει μια τέτοια προσπάθεια μέσα από μια γενική διεύθυνση Stratcom και αυτό να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για μια ποιοτική δημοσιογραφία η οποία θα εκθέτει αυτή την χειραγώγηση που μας απειλεί. Να, για παράδειγμα. Ξέρετε, εκτός Πολωνίας υπήρξε ενημέρωση από το Σπούτνικ σε σχέση με το... Τι, τι συζητάμε εδώ στο Κοινοβούλιο, στην ε, ομάδα μας και ανέφεραν και το όνομα κάποιου εμπειρογνώμονα. Ε, αυτό ήταν μια είδηση που την αντέγραψαν πολλά ΜΜΕ. Δεν ανέφεραν την πηγή, δεν ανέφεραν τα ονόματα. Να, πώς διαδίδονται οι ειδήσει και πώς η χειραγώγηση ε, εντείνεται. Μιλάμε για δίκτυα, δεν πρόκειται για μοναδική πηγή. Φυσικά και το Σπουτνίκ δεν έχει ακροατήριο εκατομμυρίων, αλλά οι ειδήσει που μεταδίδει ε, μεταδίδονται, ε, γίνονται τους πάντων αναμεταδίδονται από άλλα ε. Τέλος πάντων, να δούμε το timing τώρα για τη συνέχεια, να το με την γραμματεία. Σας παρακαλώ πάντως να κανονίσετε να ψηφίσουμε και επιψηφίσουμε την έκθεση το συντομότερο. Νομίζω ότι υπάρχει συνέντευξη για τα περισσότερα σημεία. Και εσείς κυρία Χάρμς να δούμε ε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν ε, διατύπωση του κειμένου. Ακριβώς να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη διάκριση μεταξύ Ρωσίας και μη ε, κρατικής προπαγάνδας. Βεβαίω και να γίνει διαφοροποίηση αντιμετώπισης της μιας από την άλλη πήγη προπαγάνδας. Πάντως, Σίγουρα οπωσδήποτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε απειλή και απειλές που από παντού κατευθύνονται εναντίον μας, άσχετα από την πηγή τους. Άρα εμείς θα πρέπει να αντισταθούμε. Ακριβώς θέλω να πω ότι η κυρία Χάρμς μας είπε για την προπαγάνδα στη Σκοτία. Είμαστε πολιτικοί και άρα θα πρέπει να μπορούμε και να δούμε μπροστά, να προλάβουμε τις εξελίξεις, γιατί πρόκειται για μεγάλο κίνδυνο. Επομένως, τώρα είναι η ώρα να επιδείξουμε ενότητα. Να βρούμε τις απαντήσεις. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει αυτή την έκθεση να την εγκρίνει. Και αυτό θα είναι η σωστή απάντηση σε όλες αυτές τις απειλές. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φωτίγκα λέει ο πρόεδρος. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι θα ψηφίσουμε στις 30 Αυγούστου στην Επιτροπή μας. Και να δούμε όταν φτάσει αυτή η μέρα που πέφτει Τρίτη να δούμε τι θα προκύψει. Είναι η τελευταία Τρίτη του Αυγούστου. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα στην εμερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση της ανατεθήσας από την ΑΦΕΤ μελέτης με θέμα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική σε περιφερειακό πλαίσιο. Καλώς ορίζω εδώ για το επόμενο θέμα, τον κύριο Κέραν Στάνκ, που είναι ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μελετών στο Παρίσι και έχει αναλάβει την μελέτη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μοιραστεί έτσι εκ των προτέρων η μελέτη αυτή στα μέλη μας. Καλώς ήρθατε κύριε Στάνκ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την μελέτη μας. Η πολιτική όσον αφορά την Αρκτική σε περιφερειακό επίπεδο αποτελείται από διάφορα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μας απέναντι στην Αρκτική. Έρχεται Λίγο μετά μια πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΠΑ της εκπροσώπου για την Αρκτική που αυτή έγινε σε αρχές της χρονιάς. Θα σας πω γιατί πράγματα θα σας μιλήσω. Το εύρος εφαρμογής της μελέτης. Θα μιλήσω λίγο για την Αρκτική για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά την Αρκτική. Θα αναφερθώ μετά σε διάφορες κυβερνητικές προκλήσεις στην περιοχή και τέλος θα αναφερθώ στα θέματα ασφάλειας και ενέργειας που έχουν να κάνουν με την Αρκτική και στα συμπεράσματά μου θα αναφέρω κάποιες συστάσεις. Κάποια στοιχεία κλειδί τώρα που αξίζουν τον κόπο να αναφερθούν για την Αρκτική. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα και σίγουρα θα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, διότι οποιαδήποτε καταστροφή εκεί επηρεάζει, και συνέπειε στον πληθυσμό τον ε, τοπικό και στο κλίμα γενικότερα. Η τάση είναι η μείωση τιμών το πετρέλαιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια ένα γεγονό το οποίο είχε τεράστιες συνέπειε. Το 2014 καταρχήν πέσαν οι τιμέ και αυτό είχε επιπτώσεις. Πολλέ ελπίδε δημιουργήθηκαν για το κατά πόσο στην Αρκτική θα μπορούσαμε να είχαμε ευθυνό πετρέλαιο, αυτά το 2014 πριν πέσουν οι τιμές και μετά βέβαια όταν πέσαν οι τιμές τότε πολλοί αποσύρθηκαν από τι ιδέες αυτές και τα σχέδια που είχαν για παρέμβαση στην Αρκτική. Δημογραφικά επίσης το ρωσικό κομμάτι που έτσι καλώς τη μισή Αρκτική καλύπτει η Ρωσία. Μειώνεται ο πληθυσμός εκεί. Δεν συμβαίνει το, δεν συμβαίνει το ίδιο στη Βόρεια Αμερική, όπου εκεί ο πληθυσμός είναι πιο σταθερός. Είναι 0,1% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Πάντως υπάρχει και ένα ζήτημα αστικοποίησης των πληθυσμών εκεί. Κάτι το οποίο θα μας απασχολεί σίγουρα μακροπρόθεσμα. Και βέβαια οι κλιματικές αλλαγές, οι επιπτώσεις στο κλίμα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι αλλάζει η τοπική διακυβέρνηση το Ευρωπαϊκό Τμήμα, τα κοινοβούλια των Σάμι και στον Καναδά, η Κίγριλανδία ε, τονίζουν τις δυνατότητες που έχουν ώστε να ακούγεται περισσότερο η φωνή των τόπιων πληθυσμών. Και έτσι φτάνω στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διάφορες ακτικές χώρες έχουν τη δικιά τους πολιτική. Εδώ και 30 και 20 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η πολιτική για την ακτική. Αυτό όμως τώρα αλλάζει. Βέβαια υπάρχει και κάποια συνέχεια γιατί και σε 30 και σε 50 χρόνια θα εξακολουθούμε να μιλάμε για αυτή την πολιτική. Δεν υπάρχει μόνο καταστροφή. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την Ο νέος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που διαμορφώνεται. Με την Κομισιόν, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζητάμε για την πολιτική αυτή. Υπάρχουν πολλά σχέδια που χρηματοδοτούνται. Υπάρχει μια συνέχεια στις προτερότητες κλειδί όσον αφορά την περιοχή αυτή και οι προτερότητες αυτές είναι κοινέ μεταξύ των ε, χωρών στην Αρκτική, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία, αλλά είναι κοινέ και με τον Καναδά, τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Ισλανδία, την Ορβηγία και την Ρωσία. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της αηφόρου ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας. Επαναλαμβάνονται αυτά ξανά και ξανά όταν ο Καναδάς, οι Ηνωμένε Πολιτείε προείδρευαν τα τελευταία χρόνια ε, στο Αρκτικό Συμβούλιο, αυτά επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά. Οπότε είναι θέματα κοινά για συνεργασία, κάτι το οποίο δεν μας εκπλήσει. Γιατί είναι η περιοχή μοντέλο, παράδειγμα για συνεργασία, διεθνή συνεργασία. Τώρα για τον ρόλο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρκτικές ευρωπαϊκές χώρες και άλλες έχουν στηρίξει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική. Βέβαια, κάποιες συγκεκριμένες χώρες ασχολούνται περισσότερο με θέματα ε, στρατηγικής και έχουν συζητήσει στα κοινοβούλια τους όσον αφορά τις ανακοινώσεις της Επιτροπής. Την τελευταία δεκαετία η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Λισαβόνα έχει αλλάξει. Η αρκτική πολιτική διαμορφώνεται. Είναι βέβαια πολύ νωρίς. Αλλά πάντα υπάρχει ευκαιρία να γίνουν περισσότερα. Το στοιχείο κλειδί για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική είναι το Αρκτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 8 αρκτικές χώρες, εκπροσωπούνται έξι αυτόχθονοι πληθυσμοί και παρατηρητής. παρατηρητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει να είναι παρατηρητής πριν από αρκετά χρόνια. Δεν έγινε εξαιτία κάποιων διενέξεων με τον Καναδά όσον αφορά το εμπόριο το δεξίδιο του άνθρακα. Τώρα φαίνεται ότι η Ρωσία είναι αυτή που δεν δέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητή στο Αρκτικό αυτό Συμβούλιο. Πάντως γενικά η διακυβέρνηση στην Αρκτική είναι αρκετά περίπλοκο ζήτημα, αλλά και πιο επιτυχές από ό,τι θα φανταζόταν κανείς, δεδομένου ότι θεωρείται γενικά ότι είναι ένας κενός χώρος διακυβέρνητος. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό δεν είχε γεωστρατηγική ταυτότητα μέχρι τώρα η περιοχή, μέχρι και μετά τον ψυχρό πόλεμο. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες Το Αρκτικό Συμβούλιο, όπως σας είπα, με πέντε χώρες που φτάνουν στον Αρκτικό ωκεανό, πρωταγωνιστούν. Είναι μια τύπη ομάδα προς το παρόν υπάρχουν και διάφορα περιφερειακά πλαίσια στα οποία συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και συνεργασία διασυνοριακά και με τη Ρωσία και με την Νορβηγία και με την Ισλανδία. Πολλά διαφορετικά πλαίσια συνεργασία. Η συνεργασία έχει να κάνει κυρίω με το περιβάλλον όπως φαντάζεστε, με την κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη είναι μια πολυεπίπεδη κυβερνητική συνεργασία που κατηγορούν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συζητιώνται και για στρατηγικά θέματα, στρατηγικής πιο πολύ αυτά συζητιώνται άτυπα μεταξύ των πέντε αρκτικών χωρών. Γενικά στο Συμβούλιο το Αρκτικό δεν συζητιώνται θέματα ασφάλειας. Το θέμα της ασφάλειας λοιπόν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η ίδια η είπατε, πρόσωπος είπε ότι η Αρκτική είναι σημαντική για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Όπως σας είπα, είναι μοντέλο καλής συνεργασίας η περιοχή αυτή στο κόσμο και πολλοί θα θέλανε να το αντιγράψουν αυτό το μοντέλο. Πάντα όμως δυνητικά μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Κυρίως επειδή σας είπα ότι η Ρωσία είναι μεγάλος παίκτη στην Αρκτική. Πάντως, τα μοντέλα συνεργασίας έχουν δώσει προτεραιότητα στην Εθνική Κυριαρχία, Καναδάς, Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία. Λένε, το θέμα είναι αυτό, εμείς το εξετάζουμε, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε θέματα ασφάλειας μεταξύ μας. Αυτή είναι η τάση γενικά. και αυτό και βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε όσον αφορά την διακυβέρνηση της Αρκτικής. Πρόσφατα όμως βλέπουμε ότι η Ρωσία αναπτύσσει περισσότερο τις στρατιωτικές της βάσεις. Περισσότερα ποινικά υποβρύχια από ό,τι στο παρελθόν και θα πρέπει να θέσει κανείς κάποια ερωτήματα για τη δυνατότητα να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο μια ε, επέκταση των γεωστρατογικών αντιπαραθέσεων έχει 8 μέλη και το, τα 7 από τα 8 έχουν επιβάλει κυρώσει στο 8. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα για τη συνεργασία στον ακτικό. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί η συνεργασία, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στην Ακτική Είναι βέβαια η δύναμη του status quo, έχουν πολλά να προστατεύσουν εκεί πέρα. Χρειάζονται τον ωκεανό για τα πυρηνικά τους υποβρύχια στη Χερσόνησο τη Κόλλα. Πρέπει λοιπόν να προασπίσουν αυτήν την περιοχή. Δεν είναι κατά ανάγκη μια επιθετική δύναμη. Αν δείτε τον χάρτη της Αρκτικής και αν δείτε που βρίσκονται οι στόχοι των στρατιωτικών ε, των στρατηγικών επιθέσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν, φυσικά βρίσκονται εκεί για τη Ρωσία. Επίση και τα τελευταία χρόνια η Ρωσία έχει υποσαρτήσει στην Κρυμαία, έχει υποστεί κυρώσει. Παρ' όλο αυτό υπήρξε πολύ μεγάλη πρόοδο για ένα κώδικ... κοινό κώδικα για την ε, Ακτική Θάλασσα, ε, μια ακτοφυλακή για την Ακτική με συνεργασία των Αμερικανών και των Ρώσων, συμφωνία για το ατομικό συμβούλιο που έχει να κάνει με τα θέματα της Αρκτικής έχουν βέβαια τα τελευταία δύο χρόνια δυσκολέψει κάπως αυτές τις προσπάθειες συνεργασίας. Εκεί λοιπόν θα σταματήσω για τη Ρωσία και τα θέματα ασφάλειας. Άλλες συζητήσεις για την ασφάλεια εμπλέκουν θέματα ασφάλειας του περιβάλλοντος, ανθρώπινης ασφάλειας και η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτά τα θέματα έχουν κάποια χρησιμότητα σε ορισμένες περιπτώσεις. Η Αρκτική αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια αναπτυγμένων χωρών, όπου και η ασφάλεια, η ανθρώπινη ασφάλεια δεν τίθεται με τους ίδιους όρους και όταν συζητώ για την πολιτική της Ευρώπης στιάζουμε εστιάζουμε πολύ στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή, στη συνεργασία, στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι πτυχές της ασφάλειας του περιβάλλοντος και των ανθρώπων. Και είναι χρήσιμο λοιπόν να σκεφτούμε για όλα αυτά τα θέματα. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα ασφάλειας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ε, αναδυόμενος εταίρος σε θέματα ασφάλειας. Θέλω να υπογραμμίσω τι γίνεται στο νότιο και ανατολικό τμήμα και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτά που κάνουν τα κράτη. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αυτές τις ενέργειες για την περιοχή της Ακτικής όμως, η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ειρηνική, αν εξακολουθήσει να είναι έτσι και στο μέλλον, δεν το ξέρουμε. Είναι καλύτερο λοιπόν να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, να μην περιμένουμε τα πράγματα να συνεχίσουν, να τα αντιμετωπίσουμε με τις πολιτικές μας και τις στρατηγικές μας. Ενέργεια στην Αρκτική. Και θα καταλήξω στα συμπεράσματα. Για την παραγωγή ενέργειας στην Αρκτική. Υπάρχουν φυσικά ορυκτά καύσιμα. Δεν θα υπάρξει βέβαια μαζική εξόριξη από την περιοχή της Αρκτικής. Υπάρχουν δύο σημαντικοί γείτονες, η Ρωσία και η Νορβηγία, που δίνουν σημαντικά, σημαντικές ε, ποσότητες πετρελαίου στην Ευρώπη. Για την περίπτωση της ε, Ρωσίας ε, προέρχεται και από περιοχές της Αρκτικής και για την Νορβηγία γίνεται περισσότερη ανάπτυξη περιοχών αυτών. Ε, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο με διαφορετικούς τρόπους και όχι μονάχα με την ε, χρήση αγωγών φυσικού αερίου. Μπορεί λοιπόν με την ε, ε, υγροποίηση του φυσικού αερίου να τύχει εκμετάλλευση σε αυτό το φυσικό αέριο. Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θα συνεχίσει παρά το γεγονός ότι θέλουμε να έχουμε μια οικονομία απανθρακωμένη. Δεν είναι η λύση λοιπόν η φυσική πόλη της Ακτικής ή έστω ένα σημαντικό στοιχείο συστατικό της επίλυσης των ενεργειακών μας προβλημάτων, αλλά μπορούν να είναι τμήμα της λύσης η διαφοροποίηση και η εταιρική σχέση με τις Ακτικές. Αυτές χώρες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να συζητάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε σχέση με τις πράσινες και ψυχρές τεχνολογίες, την καλύτερη χρήση ενεργειακών πόρων, διάφορους ενεργειακούς πόρους που θα συμπληρώσουν αυτούς που έχουμε τώρα πέραν των ε, υδρογοναθάκων. Μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια στα επίπεδα της ε, ζήτησης για αυτά τα προϊόντα. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε γιατί ακόμα μέσα στην στρατηγική από ανθρακοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Μπορεί κάποιε χώρε να θέλουν να επενδύσουμε περισσότερο στην εξόριξη στο, στην περιοχή της Αρκτικής, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας σε υδρογονάνθρακες και πηγές ενέργειας. Κάποια πράγματα λοιπόν πρέπει να συνεχίσει να σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή της Ακτικής. Πρώτα, και αυτό που έλαβατε στις υφιστάμενες πολιτικές, αλλά πρέπει να το επαναλάβουμε, είναι η εστίαση στις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή σήμερα, από οικονομική έποψη και από έποψη διακυβέρνησης, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ακτική και στο έδαφος των εταίρων μας σε ό,τι αφορά επένδυση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη. Πολλά τμήματα της ακτικής οικονομίας βασίζονται στην ανάπτυξη των ε, φυσικών πόρων της περιοχής και χρειάζεται και βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα αποτελέσει τον, τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας σε επίπεδο διακυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σημαντική δύναμη <clears throat> για την μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή και κυριοποίηση των ε, πόρων και της οικονομίας και μπορεί να προωθήσει την διάφανη αυτή συμμετοχή και την διαβούλευση. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα ρόλο ηγετικό σε επίπεδο περιβάλλοντος. Μπορεί να μην τους αρέσει η, και τους κατοίκους της περιοχής να τους κάνουμε κήρυγμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Καναδάς, ε, παραγωγός δεν θέλει να ακούσει για τα ευρωπαϊκά παραδείγματα. Είναι πολύ καλύτερη η δική του εμπειρία. Αλλά μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα ρόλο ως ε, ηγέτης, να δίνει τον τόνο στις διεθνείς ε, συζητήσεις με ένα τέτοιο τρόπο όμω που να μας ακούει και η άλλη πλευρά. Φυσικά, ε, οι συνήθειες του παρελθόντος παραμένουν. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε τα θέματα της ασφάλειας για την ενεργειακή προμήθεια στην ατζέντα, στο προσκήνιο της ατζέντα θέλουμε να είναι ανοιχτή, πράσινη και ειρηνική, αρκτική και θα πρέπει να εστιάσουμε στο να το επιτύχουμε και ζητώ μεγαλύτερη συνεργασία και πολιτική συνοχή μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών. Είναι νέος χώρος πολιτικής η και είναι καλό να συνειδητοποιήσουμε και περισσότερους για τα θέματα Θα Έχουμε ξεκινήσει καλά λοιπόν. Thank you very much and um, by the pronunciation of the word about I, uh, I take... Ε, έτσι όπως το είπατε το ε, about, κατάλαβα ότι έχετε καναδική προφορά, έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, συμπαθάτε με. Τώρα, ερωτήσεις. Ποιος θέλει να ρωτήσει, παρακαλώ να είστε σύντομες ερωτήσεις και παρατηρήσεις, γιατί ήδη έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με το διάγραμμα, για κονσάρι. Ευχαριστώ πολύ για την τόσο ευρία εμβριθή σας παρουσίαση η Κίνα είχε αναπτύξει δραστηριότητα και θέλανε να έχουν αρκτική χωρίς πάγους λέγανε. Τι γίνεται τώρα, γιατί όπως ξέρουμε παντού έχει αναπτύξει δραστηριότητα η Κίνα. Τι, τώρα έχουν σταματήσει να σου λένε και την άφησαν για μας. Επίσης, τι γίνεται όσον αφορά την διακυβέρνηση όσον αφορά την άσκηση μιας πολιτικής για την Αρκτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε και το περίφημο που είχε πει ο Κίσινγκερ. Ποιος ασχολείται στην ε, Επιτροπή με την Αρκτική, ποιο είναι το τηλέφωνο του. Επίσης, για πέστε μου. Τι γίνεται με τη Ρωσία, αν σας κατάλαβα καλά. Λέτε ότι η Ρωσία φέρεται επικοδομητικά για την εκδική. Συνεργάζονται με Νορβηγία, με τον ΝΑΤΟ γενικότερα. Για ποιο λόγο έχει αυτή τη στάση και συμπεριφορά η Ρωσία. And um, Mrs. Lösing, please. Κυρία Lösing. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. εντάξει, με ακούτε. Σας ευχαριστώ για την τόσο πλήρη παρουσίασή σας. Ήδη οι θερμοκρασίες σε αυτό το δωμάτιο προσεγγίζουν αυτής, αυτές τις ε, Αρκτικής και έχουμε ένα γεγονός πολυμέσων επομένως σε αυτή την αίθουσα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε κάποια σχόλια για την προβληματική του περιβάλλοντος, για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της ακτική. και επίσης να σταθείτε και στα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν και από τη μεγαλύτερη χρήση της ε, ακτική από την εμπορική ναυτιλία Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ένα πρόβλημα που είδαμε και σε περιοχές όπως η, Μολδαβία. Αλλά στην περίπτωση της Αρκτικής είναι πολύ περισσότερο ευάλωτη η φυσική ισορροπία στην ε, Ακτική και επομένως μπορούν να προκύψουν σημαντικές ε, ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και λόγω της πολυπλοκότητας του οικολογικού πλαισίου της γης μπορεί μια αλλαγή του κλίματος ή των συνδικών στην Αττική να έχουν επιπτώσεις σε ευρύτερο επίπεδο. Χαίρομαι λοιπόν που εξετάζετε αυτήν την προβληματική στη μελέτη σας και της δίνετε ιδιαίτερη έμφαση. Θα ήθελα επίσης να ξέρω ποια είναι η άποψή σας αν θα μπορούσε να υπάρξει και μία σύμβαση όπως η σύμβαση της Αρκτικής, μία σύμβαση η οποία θα αποκλείσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ασκήσεις στην Ακτική, δηλαδή θα εφαρμόσει ένα μορατόριο, και ένα, στην εκμετάλλευση των εδαφών της Αρκτικής. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο, μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι σημαντική, να είναι εφικτή και φυσικά αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο συνάδει με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης για τα θέματα της πολιτικής ασφάλειας. Αναφερθήκατε στο ρόλο της Ρωσίας στα πλαίσια αυτά και είπατε ότι παρά την επιδείνωση των σχέσεων μας με τη Ρωσία, στην περιοχή της Ακτικής εξακολουθούμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την ε, Ρωσία ότι ακόμα και η κρίση της Ουκρανίας δεν έχει, ε, δεν έχει επιδεινώσει τις συνθήκες αυτής της συνεργασίας. Αλλά συγχρόνως λέτε για τις αυξανόμενες στρατιωτικές δραστηριότητες της, ε, στην περιοχή με ιδιαίτερη εστίαση στη Ρωσία, αν το καταλαβαίνω αυτό, επικρίνεται αυτήν την στάση της Ρωσίας ή τουλάχιστον τη θεωρείται προβληματική. Αλλά δεν θεωρείται ότι οι ενέργειες χωρών του ΝΑΤΟ όπως ο Καναδάς δεν αποτελούν προβλήματα για την περιοχή. Οι στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται από άλλες χώρες εκεί δεν είναι τμήμα αυτής της προβληματικής για σας ή δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν προκλήσεις για την περιοχή της Αρκτικής. Και πάλι σας ρωτώ πώς, πώς βλέπετε τις ε, ενέργειες του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνα το 2013 και δεν μιλάω για τι ΗΠΑ σα σύνορο, αλλά μόνο του Υπουργείου Άμυνα του. Ευχαριστώ κύριε Λόζινγκ. και Μπατσίτη. Ε, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η Αρκτική παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η δε τήξη των πάγων θα έχει επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους. Ε, e, Και βέβαια άλλοι τα υπολογίζουν διαφορετικά από άλλους. Δηλαδή λέμε ότι έχουμε εκεί αυτές τις πέντε εμπλεκόμενες χώρες. Υπάρχουν εκεί πολύ πλούσιοι πόροι και αυτές οι πέντε χώρες επομένω δεν αφήνουν άλλους να αντλήσουν πληροφορίες. Μας είπατε ότι ε, ε, τα έχουν βρει αυτές οι πέντε χώρες και έτσι διαχειρίζονται και διακυβερνούν. Τι γίνεται με τη Ρωσία. Εκεί αναπτύσσει ένοπλες δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις η Ρωσία και ο στόχος είναι σαφής. Θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Υπάρχουν και στρατηγικοί στόχοι σε σχέση με την Αρκτική και για αυτό και αυξάνει. Ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία. Άρα για πέστε μας. Είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Έχουν όλοι τόσο αγαστές σχέσεις αυτοί οι πέντε. Μήπως στο μέλλον θα πρέπει περισσότερο να προσέξουμε να προσέξουμε τι προβλήματα για την ασφάλεια εγκυμονεί η περιοχή. Thank you very much. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος. Έχω μια τελευταία ερώτηση, σύντομη εγώ, κύριε Στάν. Πριν την ε, κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου, έλεγαν πολλές πηγές, πολλές εκθέσεις ότι προσέχει ενδιαφέρον η περιοχή σε σχέση με την εξόριξη, την άντληση πετρελαίου τέλος πάντων. Τώρα όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές έχουν αποσυρθεί. Ετηρούν λοιπόν, στάση αναμονή για να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου. Ε, τι έγινε, μήπως υπάρχουν και άλλες μεταβλητές, μήπως γι' αυτό παρετήθηκαν και έκαναν πίσω όσον αφορά το ενεργειακό. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ξεκινάω από το τέλος όσον αφορά επομένως αυτούς του πρωταγωνιστές του ενεργειακού. Στην Φόρεια Αμερική και στην Αλάσκα όλοι έκαναν πίσω και σταμάτησαν ε, τις δραστηριότητες όπως και οι Ρεψόλ σταμάτησαν να έχουν αυτές όλες τις ε, θαλάσσιες πλατφόρμες εξόριξης κλπ. Στην δε Ρωσία βεβαίως έχουν αποθαρρυνθεί και από τις κυρώσεις και από την ε, χαμηλή τιμή του πετρελαίου. Δεν έχουν πρόσβαση και στη δυτική τεχνολογία. Αυτό τους έχει περιορίσει. Επίσης βέβαια όντως ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Αλλά βέβαια είναι κοινή λογική ποια είναι τα, τα κριτήρια να πτύξει κανείς ε, δραστηριότητα αν θέλει να συνεργαστεί κανένα ε, με την Κίνα όταν δεν συμμετέχουν δυτικοί, αν θα το πάει στην ε, εξόριξη ε, υγροποιημένου αερίου. Τέλος πάντων, είπαμε ότι συμμετέχουν στο Αρκτικό Συμβούλιο, οι Ρώσοι, αλλά έχουμε και άλλους παρατηρητές, τους Ρώσου. Και ενδιαφέρονται γιατί από εκεί περνάει ο δρόμος προς την Ρωσία. Υπάρχει αυτός ο θαλάσσιος διάβλος και ξανοίγονται επίσης θαλάσσιες διαδρομές πιο πολύ από όσο φαντάζεται ο κόσμος, άρα υπάρχει ε, δραστηριότητα τέτοιου είδους θαλασσίων μεταφορών. Να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον πάντως ε, σε μεγάλο βαθμό ε, έχουν έντονη παρουσία, αλλά δεν είναι και πρώτος προτεραιότητα. Όμως μπορούν όντως να επιδιώκουν πολλούς στόχους ταυτόχρονα, που δεν ίσχυε αυτό πριν από 10 χρόνια. Γιατί το ρίχνανε περισσότερο στις βασικές προτεραιότητες και τίποτα άλλο. Τώρα τι γίνεται, τι προοπτικές υπάρχουν. Ε, έχουμε διμερείς επαφές έχουμε συγκεκριμένη θεματολογία. Περιβάλλον, ας πούμε, ενέργεια κλπ. Οπότε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντίστοιχα διαφορετικές οι υπηρεσίες. Έχουμε και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, άρα εξαρτάται από το θέμα. Δεν υπάρχει ένας μόνο που να ασχολείται να τον πάρετε τηλέφωνο όπως είπατε. Τώρα, γιατί είναι συνεργάτη με η Ρωσία. Γιατί εκπροσωπεί το status quo η Ρωσία. Τα πράγματα τους πάνε καλά, πέραν των κυρώσεων. Δεν υπάρχει κάτι που να τους ενοχλεί σε αυτό το μέτωπο. Άρα, προς το παρόν δείχνουν τέτοια στάση επικοδομητική. Εμείς Επίσης, ε, έχουμε συμπεριφορά επικοδομητική. Οπότε υπάρχουν και επαφές επικοδομητικές μεταξύ στρατιωτικών. Από το 2014 ξεκίνησε αυτό. Τώρα για το περιβάλλον. Ναι, δεν σας τόνισα τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων αυτών στο περιβάλλον, αλλά είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα κράτη τα οποία εκεί ε, δρούν. Γιατί η περιοχή είναι αρκετά ευάλωτη από πλευρά περιβάλλοντος. Είναι σοβαρό το θέμα. Τα πάντα είναι αβέβαια, δεν ξέρει κανείς. Εάν προχωρήσουμε σε διάφορες δραστηριότητε, ε, ας πούμε για πετρέλαιο, για ναυσιπλοεία κλπ. Δεν, δεν φαντάζεται, δεν ξέρει κανείς ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των περιβάλλων. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς θα έχουμε βιώσει μια ανάπτυξη. Τώρα ποιοι άλλοι ενδιαφέρονται, όχι κανείς πλην των αρκτικών πρωταγωνιστών. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για κάποια άλλη ρύθμιση, κάποια συνθήκη. Δεν ε, τους ενδιαφέρει. Άρα το να αλλάξει κάτι στην θεσμική ρύθμιση τους βρίσκει αντίθετος. Οι Αμερικανοί επίσης θεωρούν ότι πρόκειται για σημαντική περιοχή στρατηγικά, για πυράβλους, αλλά δεν ε, την έχουν σε υψίστη προτεραιότητα την Αρκτική πέραν ε, της περιοχής της Αλάσκας. Φιλανδία, Νορβηγία, είναι η Ευρωπαϊκή Αρκτική, ε, θετική και εκεί υπάρχει συνεργασία σε αρκτικό επίπεδο. Τώρα, τώρα έχει δημιουργηθεί ένα μικρό πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι αυτό θα εκνευρίσει την Ρωσία αν το ΝΑΤΟ αναπτύσσει κάποιες δραστηριότητε. Και για να δούμε. Πόσα θέματα έχουμε τώρα στην Αρκτική. Αυτό είναι ένα θέμα όπου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων μεταξύ των χωρών των Αρκτικών φτάνουν αρκετά προς το βορρά μέχρι να φτάσουν σε ένα σημείο που υπάρχουν αμφισβητήσεις. Είναι τόσο βόρεια οι αμφισβητούμενες περιοχές οι οποίες, ώστε για αιώνες δεν θα είναι προσβάσιμες. Μέχρι τότε θα έχουμε σταματήσει την εξάρτηση από τον άνθρακα, ελπίζω. Οπότε δεν θα χρειάζεται να ψάχνουμε για άνθρακες εκεί. Στις περιοχές των χωρικών υδάτων, λοιπόν, είναι οι περιοχές αυτές είναι οι μόνε περιοχές που βρίσκονται στα χωρικά έδατα αυτών των χωρών που είναι προσβάσιμες για εξόριξη. Και σε σχέση με την ε, αντιμετώπιση της Ρωσίας από τις άλλες ακτικές δυνάμεις είπα ότι υπήρχαν και, και σημαντικές ε, ε, επαφές στο στρατιωτικό επίπεδο που έχουν σταματήσει τώρα αλλά η Ρωσία δεν είναι κάτι το μονολυθικό στην αντιμετώπιση της, μπορούν να είναι εταίροι για πολλά πράγματα. Είναι μια δύναμη του status quo. Έχουν ε, κάθε συμφέρον να συνεχίσουν στις συναντήσεις με τις άλλες 7 χώρες οι οποίες θέλουν να επιβάλλουν κυρώσεις. Έχουν μια συνεργασία που είναι εύθραυστη αλλά συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις εξαιρετικές σας παρατηρήσεις που θα μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε για την έκθεση πρωτοβουλίας μας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή, όσον αφορά την Αρκτική. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, συνεχίζουμε. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Αναβλήθηκε το επόμενο σημείο. Άρα παραμένει ένα μόνο και αυτό είναι θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά διακυβερνητικέ συμφωνίες και μη δεσμευτικά μέσα μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και κατάργηση της απόφασης 1994 του 2012. Θα συζητήσουμε λοιπόν την πρόταση αυτή τώρα και ο κύριος Κούκαν έχει το λόγο, συγητής μας. Παρακαλώ κύριε Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω εκεί στη θέση του Πρόεδρου. Να επενθυμίσω ότι έχουμε να κάνουμε με την γνωμοδότηση που ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής για αποφάσεις ενημέρωσης του Μηχανισμού Ανταλλαγής Πληροφοριών όσον αφορά διακυβερνητικές συμφωνίες και μη δεσμευτικά μέσα στον τομέα της ένεργης της ενέργειας. Το συζητήσαμε αυτό πριν από αρκετό καιρό. Θα είμαι λοιπόν σύντομος και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Έχουμε πάρει 36 τροπολογίες. 9 από τον εισηγητή και 37 από τους άλλους συναδέρφους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που δείξατε ενδιαφέρον για την γνωμοδότηση αυτή. Το θέμα της διαφάνειας θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει συντονισμένες θέσεις, κυρίως στον τομέα της ασφάλειας. Επ' αυτού λοιπόν συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ότι διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της έρευνας πρέπει να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πριν υπογραφούν, Να υπάρχει δηλαδή αυτή η εξάντε αρχή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε τέτοια ε, συμφωνία και για συνεργασία γενικότερα με τις χώρες μέλη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ενημερώνουν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη δεσμευτικές ενεργειακές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα που έχω να σας αναφέρω. Και για τις τροπολογίες τώρα συγκεκριμένα, θέλω να πω ότι θα υποστηρίξω τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες πηγαίνουν προς την κατεύθυνση αυτή και έχουν να κάνουν με τα θετικά της απόφασης. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες του κύριου Πίτσουλα, για παράδειγμα, που προσθέτουν πράγματα για συμμόρφωση διακυβερνητικών συμφωνιών με θέματα ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με την αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω θα πρέπει να το προσέξει αυτό το θέμα. Όμως θέλω να ελέγξω κατά πόσο αυτό ευθυγραμμίζεται και με το θέμα συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε εκτενέστερα. Έχω και ένα πρόβλημα με την τροπολογία 21 εκ μέρους του ECR γιατί έχει να κάνει με το North Stream 2. Και καταλαβαίνω βέβαια και συμφωνώ με αυτό το οποίο ζητάει η τροπολογία. από την άλλη μεριά δεν πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα νομοθετικό κείμενο όπου θέτουμε αρχές και κανόνες. Εδώ συζητάμε με ρυθμίσεις που θέτουν αρχές και μηχανισμούς, αλλά όχι με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οπότε δεν νομίζω ότι η στο Nord Stream 2 ανήκει σε αυτό το κείμενο. Και τέλος, δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε συμβαστικές τροπολογίες προς το παρόν, διότι περισσότερες υποβληθήσεις τροπολογίες έχουν να κάνουν με διαφορετικές παραγράφους, με διαφορετικά ζητήματα και διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να βρούμε μια κοινή διατύπωση. Είναι ασύνηθες, αλλά έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά είμαι ανοιχτό να συζητήσω με τους κοιόδες συζητητές επί επιμέρους ζητημάτων που τους ενδιαφέρουν, ώστε να δούμε πού μπορούμε να καταλήξουμε. Αυτές ήταν οι εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ανεκτικότητα που δείξατε και για τον τρόπο με τον οποίο συζητήσατε με του ε, ΣΚΙΟΤ. Ο κ. Σπίτσουλα έχει τη δυνατότητα να λάβει τον λόγο τώρα από αυτού. Χωρίς μικρόφωνο Εντάξει, λειτουργεί τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Για τους λόγους που εξήγησε ο εισηγητής μας, καταρχήν δεν υπάρχει εξάντε έλεγχος για τη δυνατότητα παρακολούθησης των ε, διαπραγματεύσεων, έλλειψη νομικής ασφάλειας στους μηχανισμούς αυτούς και μηχανισμοί που δεν συνάδουν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απουσία ε, διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις εν εξελίξη. ο έλεγχος εκ των υστέρων δεν οδήγησε σε καμία αλλαγή των συμφωνιών. Γι' αυτό κατανοούμε ότι υπάρχει ανάγκη να τροποποιήσουμε τους κανόνες για να ξεπεράσουμε τις ε, ελλείψεις οι οποίες έχουν διακριβωθεί. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε καλή ανταλλαγή πληροφοριών και να εδραιώσουμε την ασφάλεια δικαίου όταν βλέπουμε ότι οι συμφωνίες δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τονίζω επίσης ότι υπάρχει ανάγκη ελέγχου και της Κομισιόν που και αυτή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν προθεσμίες λογικές για να μην τροχοπεδούνται οι διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται διαφάνεια σε ό,τι αφορά την προμήθεια των υδρογοναθράκων. Είναι πολύ σημαντικό όταν αναφερόμαστε σε το σημείο αυτό, να έχουμε και τον έλεγχο της κατάστασης ε, για τις χώρες διέλευσης να μπορούν και αυτές να έχουν πρόσβαση στην, στον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες σε προσιτές τιμές και σε καλή ποιότητα. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί μονάχα εάν υπάρχει σωστός συντονισμός των πολιτικών. Εν κατακλείεδη. Θέλω να τονίσω ότι αυτές οι συμφωνίες είναι μεγάλη σημασία και παράλληλα με την έγκριση του πακέτου αυτού μέτρων θα πρέπει να εργαστούμε για την βελτίωση της ενεργειακής μας ανεξαρτησίας και της ποιότητας των προϊόντων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτσουλα. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα είναι στις 5 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα. μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης αντιμετώπιση του ζητήματο των αναγκαστικών εκτοπίσεων, παρουσίαση τη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τι αναγκαστικέ εκτοπίσει και την ανάπτυξη και ανταλλαγή απόψεων με πυρογνώμονε.